Good morning to all of you. Please take your... Καθίστε σας παρακαλώ. Προσδεθείτε και απογειωνόμαστε. We are already in a time. Λοιπόν, ε, δεν υπολογίσαμε καλά το χρόνο των ε, συντονιστών. Έπρεπε όμως να αποφασίσουμε για τις ακροάσεις και δεν είχαμε πολύ χρόνο. Παρακαλώ λοιπόν, επειδή είμαστε ήδη αργοπορημένοι, να είσαστε σύντομοι και ακριβείς ε, όταν θα παίρνετε το λόγο έτσι ώστε να μην δυσκολέψουμε ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Παρ' όλα αυτά να σας ευχηθώ καλώς ήρθατε, καλό πρωινό. Ε, την έγκριση της ημερήσιας διάταξης ε, θα ήθελα να κάνουμε τώρα. Δεν βλέπω σχόλια, επομένως θεωρείται ε, εγκεκριμένη, πολύ ωραία. Ε, το σημείο 3 θα το αφήσω, ανακοινώσεις της Προέδρου μετά. Ε, υπό τα διάφορα θέλετε να προσθεθεί κάτι, όχι. Προχωράμε λοιπόν θα σας ε, ε, πω δύο λόγια όσον αφορά, θα σας κάνω μια ενημέρωση όσον αφορά τους, ε, τις συνεδρίες των συντονιστών. Υπάρχει ένα αίτημα όσον αφορά τους, την Frontex αποφάσισαν οι συντονιστές ε, να καλέσουν την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ ε, για γνωμοδότηση. Δεύτερον, υπάρχει αίτημα για ειδική διαδικασία έτσι ώστε ε, να αντιμετωπιστεί το special balayage, δηλαδή αυτή την, το σκούπισμα πούμε, το ξεκαθάρισμα των επιτροπών, των αναφορών συγγνώμη. εκλογή διαμεσολαβητού αποφασίσαμε να στείλουμε επιστολή στον πρόεδρό μας, κύριο Μάρτιν Σούλτς, ε, ζητώντας να γίνει ψηφοφορία το Δεκέμβριο για τον ε, διαμεσολαβητή, μια υπάρχει, μια και υπάρχει ένας υποψήφιος. Είχαμε μακρά συζήτηση όσον αφορά τον προγραμματισμό των δημοσίων ακροάσεων που θα οργανώσει η Επιτροπή μας ε, για το web portal και για άλλα πολλά συζητήθηκαν, αλλά λίγες αποφάσεις ε, ελήφθησαν. Εν πάση περιπτώσει, να δούμε τώρα τις προσυζήτηση αναφορές. Παρακαλώ. Κύριε Μαριά, έχετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε και κύριοι αδελφοί, σε σχέση με το ζήτημα των δημοσίων ακροάσεων, που θα οργανωθούν για το 2015, το ECR κατέθεσε δύο αναλυτικές προτάσεις. Η μία πρόταση αφορά τη διοργάνωση δημόσιας ακρόασης για το ζήτημα των γερμανικών πολεμικών επανορθώσεων. Ένα θέμα το οποίο απασχολεί τους πολίτες στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Πολωνία. Ένα θέμα το οποίο θεωρούμε πάρα πολύ σοβαρό και το οποίο αναπτύξαμε κατά τη διάρκεια της συζήτησης των συντονιστών. Όπως επίσης αναπτύξαμε και την πρότασή μας για την ε, αεροπορική τραγωδία στο Σμόλενσκ. Η πρότασή μας καταψηφίστηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης των συντονιστών. Εμείς δεν αποδεχόμαστε αυτή την απόφαση και θέλουμε να υπάρξει μια απόφαση της ίδιας της Επιτροπής στην Ολομέλειά της και να τοποθετηθούν τα μέλη αναλυτικά για το ζήτημα αυτό. Επομένως θεωρούμε ότι σε αυτό το σημείο κυρία Πρόεδρε θα πρέπει να μας δώσετε το λόγο να αναπτύξουμε την πρότασή μας και να μπουν όλες οι προτάσεις σε ψηφοφορία διότι θεωρούμε ότι το σώμα εν συνόλο πρέπει να αποφασίσει για αυτό το θέμα που είναι πολύ σημαντικό. Εμείς ιδίω το ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων το θεωρούμε κορυφαίο θέμα που απασχολεί την Ελλάδα αλλά και την Ιταλία και την Πολωνία και θέλουμε εδώ να τοποθετηθούν ατομικά οι συνάδελφοι και να υπάρξει ψηφοφορία και ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του. Εμείς εμένουμε στην άποψη αυτή και θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει συζήτηση και ψηφοφορία και για τις δύο προτάσεις τις οποίες υποβάλαμε για τη συζήτηση για τις γερμανικές πολεμικές επανορθώσεις και για το αεροπορικό δυστύχημα στο Σπόλενς. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε κύριε Μαριά, όντως αυτό ήταν, στο θέμα, ήταν θέμα για τους συντονιστές. Εκεί συζητήσαμε το πώς θα δουλέψουμε για τις ακροάσεις. Μαργκρέτε. Κύριε Μαριά, πολύ σύντομα. Εσείς επιμείνατε να ψηφίσουμε άμεσα και ε, οι περισσότεροι από εμά θεωρούσαμε ότι δεν είμαστε έτοιμοι για να κάνουμε αυτήν την συζήτηση και να πάρουμε αυτή την απόφαση. Γι' αυτό ζητήσαμε περισσότερο χρόνο και εσείς δεν μας τον δώσατε, δεν συμφωνήσατε με τον περισσότερο χρόνο αυτό. Ε, εάν επιμένετε, εάν επιμένετε, αφήστε με να τελειώσω. Κοιτάξτε, δεν θέλω να είμαι αγενής, αλλά εάν επιμείνετε είμαι σίγουρη ότι θα γίνει ψηφοφορία και θα καταψηφιστεί η πρότασή σας. Λοιπόν, νομίζω ότι καλό θα ήταν να μας δώσετε λίγο χρόνο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να το ξαναδούμε το θέμα, να δούμε όλα τα στοιχεία του. Βεβαίως, εάν επιμείνετε θα καταψηφίσουμε και θα τελειώνει η υπόθεση. Okay, let me put it this way. Πρόεδρος, θα προσπαθήσω να είμαι ευγενής αποφασίσαμε στους συντονιστές να κάνουμε ακρόαση για την πρωτοβουλία Ευρωπαίων πολιτών. Αποφασίστηκε αυτό, είχε ήδη ληφθεί η απόφαση. Δεύτερον, αποφασίσαμε να υποβάλουμε αίτημα για δεύτερη ακρόαση ε, για το πρώτο εξάμεινο του 2015, να, το, να υποβάλουμε το αίτημα λοιπόν στην αρχή του Κοινοβουλίου και προτείνουμε ακρόαση για το δικαίωμα υποβολής αναφοράς ε, συνδυασμένο με πληροφορία για την δεύτερη φάση του web portal. Ε, κοιτάξτε, εσείς φαίνεται ότι δεν βλέπετε τα πρόσωπα των ε, ε, συναδέλφων, αλλά εγώ διαβάζω καθαρά στα πρόσωπά τους ότι δεν υπάρχει πλειοψηφία που να στηρίζει την πρόταση αυτή που υποβάλλεται. Γι' αυτό λοιπόν είπαμε να το αφήσουμε και για την επόμενη συνεδρίαση, οπότε θα συζητήσουμε το δεύτερο τμήμα του έτους 2015 και ποιες ακροάσεις θα γίνουν εκεί. Προφανώς δεν συμφωνείτε, αλλά σας παρακαλώ να αποσαφηνίσετε τη θέση σας μία και καλή τώρα. Η θέση μου είναι σαφής. Σας ζήτησα εγώ ο ίδιος στη συνεδρία των συντονιστών να μην ληφθεί απόφαση σήμερα προκειμένου να συζητηθούν αναλυτικά όλες οι προτάσεις. Εγώ αυτή την πρόταση σας έκανα στην αρχή. Εν συνεχεία, σε επίπεδο συντονιστών επιμείνατε να υπάρξει απόφαση για το τι θα γίνει στο πρώτο εξάμεινο και θέλατε να μην μπουν σε ψηφοφορία οι προτάσεις. Γι' αυτό και ζήτησα και μπήκαν σε ψηφοφορία οι προτάσεις σε επίπεδο συντονιστών. Υπάρχει λοιπόν μια απόφαση η οποία είναι από τους συντονιστές με την οποία εγώ διαφωνώ. Τώρα επειδή όλα γίνονται ανοιχτά και δημόσια και στο φως βλέπω μια άλλη αλλαγή. Λέτε ότι δεν απερίφθη η πρότασή μου και θα τη δείτε στο δεύτερο εξάμεινο. Αυτό είναι μια διαφορετική θέση. Αν λοιπόν η πρότασή σας και η απόφασή σας είναι ότι στο δεύτερο εξάμεινο θα συζητήσουμε την πιθανότητα να γίνει συζήτηση για τις γερμανικές αποζημιώσεις και το Σμόλενσκ που σημαίνει ότι αναβάλλετε την απόφαση και δεν την έχετε απορρίψει τότε ευχαρίστως να το συζητήσουμε για το δεύτερο εξάμεινο αλλά η απόφαση που πήρατε προηγουμένως στους συντονιστές είναι να απορρίψετε την, απόφαση, την πρότασή μου. Γι' αυτό και το βάζω στο σώμα. Αν λοιπόν αποδέχεστε ότι είναι ανοιχτή η πρότασή μου για τις γερμανικές αποζημιώσεις και το αεροπορικό δυστύχημα στο Σμόλες για το Β' εξάμεινο, από εκεί και πέρα να το δούμε. This was my intention. Αυτή ήταν η πρόθεσή μου εξ αρχής. Ακριβώς αυτή ήταν η πρόθεσή μου και αυτή ήταν η απόφαση. Ίσως ήταν, είσαστε πολύ εκνευρισμένο και δεν το κατανοήσατε. Ο κύριος Μαριάς λέει ναι ξέρω ποια απόφαση ήταν που λήφθη και υπάρχουν και τα αρχεία άλλωστε τα πρακτικά τα, στα οποία μπορούμε να δούμε η πλειοψηφία α, καταψήφισε γενικώ την πρότασή μου. Τώρα εάν αποφασίσετε ότι οι προτάσεις μου είναι ανοιχτές προς συζήτηση και μπορούν να ολοκληρωθούν στο δεύτερο εξάμεινο του 2015 τότε μπορούμε να το συζητήσουμε και να το συμφωνήσουμε. Ναι μαζί με τις προτάσεις των σοσιαλιστών και δημοκρατών που έφτασαν γραπτά σήμερα το πρωί. Ωραία, ξέρω τι πρέπει να κάνουμε και πώς θα προχωρήσουμε με την επιστολή που θα στείλουμε στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου. Να προχωρήσουμε όμως τώρα. Να προχωρήσουμε στις αναφορές ε, τις οποίες ήρθατε για να συζητήσουμε. Όχι, όχι, όχι, όχι. Έχουμε πρώτα, ναι, έχετε δίκιο, μπερδεύτηκα. Έχουμε στο σημείο 6 την ετήσια έκθεση ε, και αναφορά για τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητού, ο κύριος Βαλέσα. Θα είμαι σύντομος, κυρία Πρόεδρε. Πρόκειται για μια πάρα πολύ καλή έκθεση που έκανε η ε, διαμεσολαβήτρια η κυρία Οράιλη και, νομίζω ότι ε, την είδαμε και πριν από λίγο καιρό, παρουσίασε την έκθεσή της και πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι ότι η εργασία της είναι εξαιρετική. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι η εργασία ε, αποτελεί συντονισμό, συνδυασμό της εργασίας του κυρίου Διαμαντούρου που ε, έφυγε από τη θέση αυτή πέρσι και της κυρίας οράλή που ε, ανέλαβε ως διάδοχός του το δεύτερο μισό του χρόνου. Η διαμεσολαβήτρια πραγματικά ανέλαβε άμεσα την εργασία της στις 24 Σεπτεμβρίου του 2014 ακούσαμε την παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης και θα ήθελα να την ε, συγχαρώ για την έκθεση αυτή. Είναι μια έκθεση η οποία δείχνει μεγάλο βαθμό προσβασιμότητας ε, και είναι όπως λέμε user friendly, φιλική προς το χρήστη. Ο ρόλος του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητού ε, είναι να βοηθάει τους πολίτες, να γεφυρώνει το χάσμα που υπάρχει μερικές φορές ανάμεσα στους πολίτες και τα ευρωπαϊκά ε, όργανα και πραγματικά έχει συμβάλει στο στόχο αυτό η ε, διαμεσολαβήτρια και αυτό διαφαίνεται σαφώς στην έκθεση. Ε, υπάρχει ένα σκέλος ε, της έκθεσης που αναφέρεται στην καλή διοίκηση και καλή διαχείριση. Ε, μονάχα ένα πρόβλημα έχουμε σε αυτό το κεφάλαιο, το θέμα της μετάφρασης. Θα θέλαμε η μετάφραση να γίνεται σε όλες τις γλώσσες έτσι ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό όλοι. Ελπίζουμε ότι σύντομα θα αλλάξει. 11 Νοεμβρίου θα συζητηθεί η έκθεση αυτή και ευελπιστώ ότι θα ψηφιστεί στην Επιτροπή στις αρχές Δεκεμβρίου ενώ στην Ολομέλεια θα φτάσει για ψηφοφορία τον Ιανουάριο. Ξέρω ότι είναι φιλόδοξο το πρόγραμμα αλλά αυτό το έγγραφο εργασίας είναι ήδη διαθέσιμο, ε, έχουμε πρόσβαση όλοι σε αυτό και ελπίζω ότι θα ε, επιτύχουμε αυτά τα χρονικά όρια. Θα ήθελα να ε, διαβεβαιώσω ότι είμαι ανοιχτός ε, σε σχόλια, σε οποιαδήποτε συζήτηση θα ήθελαν ε, οι συνάδελφοί μου να έχουμε. Η εργασία για, την έκθεση αυτή ε, ελπίζω ότι θα ολοκληρωθεί σε πνεύμα καλής συνεργασίας έτσι ώστε να εφαρμόσουμε βέλτιστες πρακτικές. Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Ευχαριστούμε για την εργασία σας η οποία είναι ουσιώδης ε, και πιστεύω ότι με τον τρόπο αυτό θα ενδυναμωθούν και οι δεσμοί που μας συνδέουν με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι ε, δουλέψατε πάρα πολύ καλά. Είσαστε έμπνευση για μας. Μακάρι όλοι να μπορούμε να δουλέψουμε με τον ίδιο τρόπο. Παρακαλώ κυρία Σμέτση. Um, Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Είμαι σκιώδες από μέρους των σοσιαλιστών για την έκθεση αυτή. Και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Βαλέσα για την εξαιρετική του εργασία και φυσικά ευελπιστώ ότι θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε σε άλλες εκθέσεις σαν σκιώδης εισηγητρία. Θα ήθελα παρόλα αυτά να αναφερθώ σε κάποια από τα σημεία. Βέβαια το κείμενο το πήραμε χτες το βράδυ, παρόλα αυτά το διάβασα. Όσον αφορά λοιπόν το πρώτο αυτό σχέδιο που βλέπω, κάποιες από τις ε, παραγράφους θέλουν ίσως περισσότερο, περισσότερη επεξεργασία, να προσθέσουμε κάποια σημεία. Παραδείγματο χάρη, ο Ombudsman φέτος φαίνεται ότι είχε επαφή με πάνω από 2.000 άτομα και ασχολήθηκε με 400 περιπτώσεις. Αυτό είναι κάτι που ξεπερνάει τους αριθμούς των προηγούμενων ετών. Και φυσικά, όπως είπε ο κύριος Φαλέσα, η νέα ομπούτσμαν σίγουρα εποφελήθηκε από την εμπειρία του προηγούμενου, αλλά βελτίωσε σημαντικά τα πράγματα. Τώρα, ε, το θέμα είναι αν είναι παραδεκτά ή όχι τα αιτήματα που υποβάλλονται στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Αυτό πρέπει να μας το πει γιατί πολλές φορές ε, δεν είναι παραδεκτά τα αιτήματα. Πρέπει λοιπόν να εξηγήσουμε ίσως καλύτερα στον Ευρωπαίο πολίτη πώς να έχει άμεση πρόσβαση στον Ευρωπαίο διαμεσολαβητή. Πρέπει να μειώσουμε την γραφειοκρατία, αυτό είναι δική μας δουλειά. Βλέπω παραδείγματο χάρη ότι 64% των ε, προσφυγών, των ετοιμάτων είναι κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μόνο 3% κατά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό δείχνει μία τάση και τις περισσότερες φορές βλέπουμε ότι τα κύρια θέματα που αφορούν τους Ευρωπαίους πολίτες είναι κακοδιαχείριση και έλλειψη διαφάνειας. Ολοκληρώνω, δεν θέλω να πάρω το λόγο για πολύ χρόνο. Το θέμα της υπηρεσίας Frontex. Και εδώ υπάρχουν ε, προβλήματα. Ε, κατά 20% εδώ οι αναφορές ε, αφορούν την Frontex και περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. Το θέμα TTIP επίσης, γνωρίζουμε όλοι αυτό το θέμα. Οι Ευρωπαίοι πολίτες βέβαια δεν γνωρίζουν ακριβώς τι είναι αυτή η συμφωνία TTIP. Και εδώ λοιπόν, επειδή θα επηρεάσει τις ζωές όλων μας και επειδή υπάρχει μεγάλη ανησυχία από μέρους των Ευρωπαίων πολιτών, πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε πιο διαφανείς. Παρακολουθώ λοιπόν όλα τα θέματα, συνεργάζομαι με τον εισηγητή, τον οποίον άλλη μια φορά θέλω να συγχαίρω. Thank you very much, Ευχαριστώ πολύ, Μαργκρέτα. Πιστεύω ότι καλή ιδέα θα ήταν ε, Καλό θα ήταν να το συζητήσουμε το θέμα αυτό, το είπα και στη συνεδρίαση των συντονιστών. Νομίζω ότι ολόκληρο το Κοινοβούλιο θα πρέπει να καταλάβει καλύτερα και να ενημερωθεί περισσότερο για την, τον ρόλο του διαμεσολαβητού, το τι έχει κάνει και ε, βεβαίως όλοι είναι προσκεκλημένοι όταν ε, γίνεται η ακρόαση, αλλά την προηγούμενη φορά ήταν λίγο παράλογη η κατάσταση. Δεν έγινε ε, έτσι ένα επίσημο καλωσόρισμα, δεν την είδαμε πραγματικά την κυρία Οράιλεϊ. Νομίζω ότι θα πρέπει να το κάνουμε αυτό την επόμενη φορά. Κύριε Μαριά, παρακαλώ. Ε, ε, σαν σκιώδης ήθελα να πω ότι θα συνεργαστούμε με τον κύριο Βαλέσα για να έχουμε μια πάρα πολύ καλή ε, παρουσία και μια καλή έκθεση. Βεβαίως ε, δεν είχαμε την ευκαιρία να μελετήσουμε σε βάθος την έκθεση επειδή μας διανεμήθηκε χτες αργά μετά τις 8 η ώρα και αντιλαμβάνεστε ότι όλες αυτές οι εκθέσεις χρειάζονται λίγο χρόνο για να μπορούμε να τοποθετηθούμε με σαφήνεια και με άνεση. Νομίζω όμως ότι από μια πρώτη ε, ματιά και διάβασμα το οποίο έγινε φαίνεται ότι είναι μια ισορροπημένη έκθεση η οποία αποσκοπεί στο να συμβάλλει να βγάλουμε σημαντικά συμπεράσματα να βοηθήσουμε την ε, λειτουργία του Ombudsman, του διαμεσολαβητή ο οποίος πραγματικά ε, κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και νομίζω ότι σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να πάμε και να έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε και κάποιες τροπολογίες. Δύο ζητήματα νομίζω ότι μπορώ να θίξω σε μια πρώτη φάση για να το έχουν υπόψη και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Το πρώτο ήδη υπόθηκε αφορά τη Frontex και εκεί είναι ένα σοβαρό ζήτημα διότι πάρα πολλές καταγγελίες αφορούν τη λειτουργία της Frontex η οποία ε, ενεργεί σε ένα ευαίσθητο τομέα ο οποίος έχει σχέση με τη διαφύλαξη των συνόρων αλλά βεβαίως αντιμετωπίζουν ε, τεράστιο αριθμό και προσφύγων αλλά και παρανόμων μεταναστών. Επομένως εδώ ο τρόπος λειτουργίας της Frontex είναι πράγματι ένα σημαντικό θέμα το οποίο μας απασχολεί. Και το δεύτερο έχει σχέση με με την εξωθεσμική λειτουργία της Τρόικας, το οποίο έθεσα και την προηγούμενη φορά κατά τη συζήτηση που είχαμε με την κυρία Διαμεσολαβήτρια. Δηλαδή υπάρχουν όργανα πλέον εκ των πραγμάτων που είναι η Τρόικα και που είναι δύο όργανα ουσιαστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που λειτουργούν όμως ως Τρόικα, στην ουσία είναι ένα όργανο εκτός των επισήμων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν ελέγχεται ως προς τον τρόπο λειτουργίας του, έχει πολλές μορφές κακοδιοίκησης και έλλειψης διαφάνειας, παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό λοιπόν το κομμάτι θα πρέπει σοβαρότατα να το δούμε και εμείς θα το θίξουμε στην έκθεση, διότι υπάρχουν ε, λειτουργίες της ίδιας της Επιτροπής ως μέλος της Τρόικας ή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ως μέλος της Τρόικας που έρχονται σε σύγκρουση με τη λειτουργία των οργάνων αυτών με βάση τις εντολές που έχουν από τη συνθήκη. Δηλαδή η, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι τεχνικός σύμβουλος της Τρόικας, ταυτόχρονα είναι και δανειστής ορισμένων κρατών και ταυτόχρονα πρέπει να επιτελέσει και το ρόλο της ως Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Υπάρχει λοιπόν μια σύγκρουση λειτουργιών και σύγκρουση συμφερόντων. Αυτά τα δύο ζητήματα που σας ανέφερα εμείς θα τα θίξουμε αναλυτικά. Βεβαίως στις επόμενες συνεδριάσεις θα συνεργαστούμε με τον κύριο εισηγητή, τον κύριο Βαλέσα, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι είναι κάτι και που η ίδια η διαμεσολαβήτρια στη συζήτηση που είχαμε πριν από μία εβδομάδα εδώ τα θεωρεί σημαντικά και νομίζω ότι πρέπει να ανοίξει και εκεί ένα μεγάλο κεφάλαιο ελέγχου της λειτουργίας της Τρόικας. Ευχαριστώ. Thank you. Thank you. I Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω. Α, όχι, κάποιος άλλος, η Ελεονόρα. Ο, λοιπόν, ήθελα μόνο να σας πω ότι ο σκιώδης συζητητής για το FTD δεν έχει ακόμα οριστεί, αλλά ως θα το κάνουμε. Και βεβαίως με μεγάλη ευχαρίστηση θα ε, συνεργαστούμε και εμείς για το θέμα αυτό, όπως και οι άλλοι συνάδελφοι. Ευχαριστούμε, Πεατρίς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο για αυτή την πρώτη έκθεση. Έχουμε μια θαυμάσια ευκαιρία με αυτή τη νέα Επιτροπή Αναφορών να αποδείξουμε όχι μόνο στα όργαλα και στους πολίτες ότι είμαστε διόψεις του ίδιου νομίσματος. Και αυτό το νόμισμα θα πρέπει να δουλεύει συνέχεια αρμονικά και από τις δύο όψεις. Στην έκθεση της διαμεσολαβήτριας Υπάρχει το σημαντικό σημείο διαφάνειας, όχι μόνο όσον αφορά τις εμπορικές συμφωνίες, αλλά και το φαινόμενο των περιστρεφόμενων θυρών. Από αυτή την άποψη, νομίζω ότι ακριβώς επειδή, επειδή εμείς είμαστε και το παράθυρο και η πόρτα των πολιτών στα όργανα, θα πρέπει να αποτελούμε τον κύριο συνεργάτη και προωθητή της δουλειά της διαμεσολαβήτριας. Γι' αυτό ακριβώς θα υποστηρίξω την έκθεση αυτή. Δεν έχουμε στην Άλντε συμφωνήσει επί αρχής, αλλά νομίζω ότι εγώ θα είμαι ως shadow. Τέλος, να υπογραμμίσω στα πλαίσια της έκθεσης αυτής ότι συμφωνώ απόλυτα με την πρόταση της Μαργκρέτε. Δηλαδή, να υποστηρίξουμε, να υποστηρίξουμε την ε, διαμεσολαβήτρια όταν αυτή εκλεγεί. Το θέμα ανοσίας και αν το αποδεχτούν όλα τα μέλη και όλο το κοινοβούλιο ως θέμα προάσπισης των πολιτών που και εμείς οι ίδιοι είμαστε εδώ με αυτό το ρόλο, τότε οι δράσεις της Δεμψαλαβήτριας θα έχουν περισσότερη ισχύ και αναγνώριση. Ευχαριστώ. Now, Yarek, the floor is yours again. Κύριος Βαλέσα, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους για τις συνεισφορές, τις προτάσεις σας. Κάτι που σίγουρα πρέπει να υπογραμμίσουμε είναι ότι πρόκειται για μια ετήσια έκθεση που αναφέρεται στο 2013. Μην ξεχνάτε λοιπόν ότι αυτά προετοιμάστηκαν από την κυρία Ομπουτσμαν και θα ψηφίσουμε τον Ιανουάριο, κλείσουμε δηλαδή το έτος 2013, ενώ ήδη το 2014 θα έχει ολοκληρωθεί και θα συνεχίζεται η δράση της κυρίας Όμπουτσμαν με τον ίδιο τρόπο. Θέλω να πω λοιπόν ότι πρέπει να στοχεύσουμε τα σημεία και τις προτάσεις που μας έχει υποβάλει στην έκθεσή σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα της πρόσβασης στον Ευρωπαίο Μεσολαβητή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα της διαφάνειας και τα δύο χρήζουν βελτιώσεων. Έκανε πολύ σημαντικό έργο η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια για την βελτίωση όλων αυτών των διαδικασιών. Σίγουρα η μεγαλύτερη διαφάνεια και η καλύτερη πρόσβαση είναι κάτι που δεν μπορεί παρά να βελτιώσει ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Τώρα, το θέμα Frontex. Πολύ σημαντικό. Δεν ξεχνάτε όμως ότι υπάρχει ειδική έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή που ασχολείται με την Frontex είναι κάτι που σαφώς ενδιαφέρει και την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και τη δική μας. Σημαντική έκθεση, αλλά επαναλαμβάνω ότι αυτό είναι το θέμα που θα επεξεργαστεί με πολύ περισσότερες λεπτομέρειες η άλλη έκθεση. Το θέμα τώρα του αριθμού των αναφορών, η πρόσβαση στον Ευρωπαίο διαμεσολαβητή, όταν μας παρουσίασε την έκθεσή της η διαμεσολαβήτρια, ήταν ε, σαφές το τι έκανε για να βελτιώσει τα πράγματα σε σχέση με τον προηγούμενο Ευρωπαίο διαμεσολαβητή. Υπήρχε συμφόρηση, υπήρχαν σαφώς ε, πολλές εκρεμείς περιπτώσεις και οι προσπάθειές της βελτίωσαν την κατάσταση. Θα συναντήσω λοιπόν την ε, Ευρωπαία Ομπουτσμαν στο άμεσο μέλλον και σίγουρα θεωρώ ότι με τις προτάσεις σας η έκθεσή μου θα βελτιωθεί και θα εμπλουτιστεί. Θα συνεχίσουμε λοιπόν τη συνεργασία μας. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος. Να σας δώσω και κάποιες ημερομηνίες, το χρονοδιάγραμμα. Όλες οι μεταφράσεις θα είναι διαθέσιμες στις 28 Οκτωβρίου. Στις 11 Νοεμβρίου θα εξετάσουμε το σχέδιο έκθεσης. Στις 12 Νοεμβρίου είναι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα εδώ στις 2 Δεκεμβρίου. Στην Ολομέλεια θα ψηφίσουμε τον Ιανουάριο. Διαβάστε το. Υποβάλλετε τις τροπολογίες σας και νομίζω ότι με μεγάλη γενεοδορία ο εισηγητής θα αντιμετωπίσει τις προτάσεις σας. Νομίζω ότι είναι εδώ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προχωρούμε στο σημείο 7, αναφορά 0745-2013, Γιάννης Δάρας, εξ των συντακτών τύπου Πρόκειται για τα ποσά που καλούνται να πληρώσουν στην Ευρώπη. Ο κύριος Δάρας είναι παρόν. Ο κύριος Ντέιβιτ Νέρτ είναι επίσης εδώ. Ο Ζαν Πολ Σαβάρ επίσης. Και οι τρεις σας είστε εδώ. Μπορείτε λοιπόν να πάρετε το λόγο, αλλά έχετε μόνο δύο λεπτά ο καθένας. Κύριε Δάρα. Αξιότιμε, κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σαν πρόεδρος της IPS Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αθλητικών Συντακτών που εκπροσωπεί 48 ευρωπαϊκές χώρες με 55.000 μέλη, επαγγελματίες αθλητικούς συντάκτες, σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης που εργάζονται 365 μέρες το χρόνο κάτω από δύσκολες συνθήκες. Σας ευχαριστούμε για αυτή την πρόσκληση. Τα τελευταία χρόνια ορισμένες ευρωπαϊκές αθλητικές ομοσπονδίες ή διοργανωτές αθλητικών γεγονότων έχουν δημιουργήσει τις δικές τους λίστες μέσων μαζικής ενημέρωσης και δημοσιογράφων προσπαθώντας να ελέγξουν τα μονοπάτια της πληροφόρησης. Αγωνιζόμαστε ενάντια σε αυτό το φαινόμενο το οποίο είναι αντίθετο. Πρώτον στην ελευθερία του τύπου από την πλευρά των δημοσιογράφων. Δεύτερον στο δικαίωμα της ενημέρωσης από την πλευρά των Ευρωπαίων πολιτών τρίτον στο δικαίωμα του ίσου και δίκαιου ανταγωνισμού από την πλευρά των εμπορικών και εταιρικών σχέσεων πριν είναι αργά θα πρέπει η ευρωπαϊκή ένωση να αναμειχθεί ενεργά και να απαιτήσει τον σεβασμό των θεμελιωδών αρχών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των αποφάσεων κανονισμών και οδηγιών και αν χρειαστεί να ψηφίσει νέου. σίγουρα μπορούν να υπάρχουν αποκλειστικά εμπορικά δικαιώματα για τις ραδιοφωνικές μεταδόσεις αθλητικών γεγονότων αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να απαιτούνται χρήματα για διαπιστεύσει ή να τίθενται περιορισμοί για τι συνεντεύξει τύπου πριν ή μετά τα αθλητικά γεγονότα ή για δηλώσεις στη λεγόμενη μεικτή ζώνη από τους αθλητές. Μέσα στα όρια που μας επιτρέπει ο νόμος δεν μπορούμε να δεχθούμε αυθαιρεσίες από συλλόγου, ομοσπονδίες ή οργανωτών αγώνων. Στην ουσία μιλάμε για εμπορικές εταιρείες που έχουν την μορφή των συλλόγων, clubs, που αποφασίζουν ποιοι ραδιοφωνικοί σταθμοί θα πληρώσουν και ποιοι όχι αυτός είναι και ο λόγος της αναφοράς μας και ως πρόεδρος της IPS Europe θα υπερασπιστώ τα δικαιώματά μας. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο David Ναέρτ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της IPS Europe και πρόεδρο των Βέλγων Αθλητικών Συντακτών και στον κύριο Ζαν Πολ Σαβάρ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της IPS, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, για να σας παρουσιάσουν ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα και να σας δείξουν πόσο επικίνδυνα διωγγώνεται και καθημερινά το πρόβλημα αυτό. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ εγώ. Now the floor goes to Mr. Nart. Ο κύριος Νάρτ, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα να δώσω κάποια παραδείγματα προβλημάτων και δυσκολιών. Το 2011 στην αντιπαράθεση Manchester United Μασαλία είδαμε ότι δεν υπήρξαν προβλήματα στον πρώτον αγώνα. Αντίθετα, 26.000 ευρώ ζητήθηκαν για τον δεύτερο αγώνα, κάτι που δεν μπορεί να πληρώσει απολύτω κανένα ραδιοφωνικό σταθμός, με αποτέλεσμα στη Γαλλία να μην αναμεταδοθεί ο αγώνας. Είδαμε ότι η UEFA επιτρέπει να υπάρχουν εταιρικές σχέσεις μεταξύ των αθλητικών συλλόγων και κάποιων ε, σταθμών με ένα συγκεκριμένο ποσό που δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 1000 ευρώ. Είδαμε όμως παραδείγματο χάρη ότι ένας Ρουμανικό ραδιοφωνικός σταθμός αναγκάστηκε να πληρώσει πάνω από 4.000 για την αναμετάδοση ενός αγώνα με το, την ομάδα του Βουκουρεστίου. Βλέπετε ότι τελικά ο κάθε σύλλογος αθλητικός πρέπει να αποφασίσει ποιο θα είναι το μέσο που θα αναμεταδώσει τον αγώνα. 17 εκατομμύρια ευρώ πλέον ζητούν ε, από την για την αναμετάδοση των αγώνων στη Λίγκα. Μα πρόκειται για ποσά τα οποία όπως καταλαβαίνετε είναι υπερβολικά υψηλά. Και υπάρχουν και πολλά άλλα παραδείγματα. Παραδείγματος χάρη στους ποδηλατικούς αγώνες, βλέπουμε την Παγκόσμια Ομοσπονδία να ζητά 250 ευρώ, αλλιώς δεν μπορούσαμε να καλύψουμε τους ποδηλατικούς αγώνες. Ευχαριστώ πολύ. Ο Ζων Πολ Σαβάρ έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, Βεβαίως όλα αυτά είναι αθλητικά γεγονότα. Παρ' όλα αυτά θεωρούμε ότι θα πρέπει να προστατεύσουμε την ενημέρωση στον τομέα του αθλητισμού. Θα πρέπει να ισχύει εδώ ο χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει άμεση και δωρεάν πρόσβαση για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όπως εμείς ερχόμαστε εδώ και μπορούμε δωρεάν να έχουμε άμεση πρόσβαση στην Επιτροπή σας. Στη Γαλλία αυτό ισχύει, γιατί εμείς έχουμε συμφωνήσει με τους πολιτικούς των χωρών μας και έχουμε τον ε, νόμο ε, του Υπουργού Λαμούρ που τηρείται τελικά στη Γαλλία από το σύνολο του τομέα. Το ίδιο και από τους ε, αλλοδαπούς που έρχονται στην Γαλλία για να οργανώσουν παγκόσμια πρωταθλήματα, όπως του ράγμπι παραδείγματο χάρη. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ράγμπι θέλησε να ζητήσει από τα μέσα για την αναμετάδοση. Θεώρησε παραδείγματο χάρη ότι μπορεί να απαγορεύεται η πληρωμή από μέρους των γαλλικών ραδιοφωνικών σταθμών. Προσπάθησε όμως να κάνει κάτι τέτοιο με τους ξένους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Αυτό απαγορεύεται στη Γαλλία. Και το παράδειγμα του αγώνα Μάντσεστερ Μασαλίας και τα 26.000 ευρώ που ζητήθηκαν ήταν παράνομα. Εγώ λοιπόν ζήτησα από τους συναδέλφους να προετοιμάσουν αυτή την αναφορά. Κύριε Πρόεδρε, εγώ είμαι υπέρμαχος της Ευρώπης πιστεύω στην Ευρώπη και θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να προστατεύσουμε βάσει κανόνων και με νομοθεσία στην Ευρώπη για να προστατεύσουμε αυτόν τον τομέα. Αυτό που συμβαίνει αλλού στον κόσμο είναι πολύ χειρότερο από αυτά που συμβαίνουν στην Ευρώπη. Πρέπει να προστατεύσουμε λοιπόν τον αθλητισμό. Εμείς βεβαίως δεχόμαστε το οικονομικό κομμάτι του αθλητισμού, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτά τα ακραία φαινόμενα τα οποία αποκλείουν τους ε, φτωχότερους από τον αθλητισμό. Βλέπετε ότι αν κάποιος αγοράσει, παραδείγματος χάρη ένα προϊόν, πρέπει να το πουλήσει. Δεν είναι δυνατόν ένας ε, διευθυντής ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού καναλιού ο οποίος έχει πληρώσει ακριβά την αναμετάδοση ενός γεγονότος να πει κατόπιν στους δημοσιογράφους αυτό το προϊόν δεν αξίζει τίποτα, θα το δώσουμε δωρεάν. Δεν είναι δυνατόν. Θα πρέπει λοιπόν πραγματικά οι δημοσιογράφοι να διατηρήσουν την ανεξαρτησία τους βάσει της χάρτας των δικαιωμάτων. Κυρία Πρόεδρε, δεν έχω πλέον χρόνο. Ελπίζω να καταλάβατε αυτά που ήθελα να σας πω. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα το λόγο έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κύριος Σαντόριο Μάκλεν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα υπενθυμίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ε, η ανάμειξη που μπορεί να έχει όσον αφορά τον αθλητισμό είναι η προώθηση του αθλητισμού. Δυστυχώ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να διερευνήσει τη συμμόρφωση ε, των ομοσπονδιών ή άλλων αθλητικών οργανισμών ε, με ε, όργανα ή εργαλεία όπως είναι η Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ή παρόμοιες παρομοιες συνθηκε όσον αφορά τον χάρτη θεμελιδών δικαιωμάτων. Είναι ε, σαφές ε, ότι υπάρχει και προβλέπεται στο άρθρο 11 η ελευθερία του τύπου. Παρόλα αυτά δεν είναι δυνατόν και δεν μας επιτρέπεται οποιαδήποτε παρέμβαση ενώπιον δημοσίων αρχών υπενθυμίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι οι διατάξει ε, τη χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ε, ε, αναφέρεται και στις αρχές της επικουρικότητας, αλλά μόνο εφόσον εφαρμόζεται ενωσιακός νόμος, πράγμα που δεν ισχύει στην προκείμενη περίπτωση. Επομένως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι σε θέση να ξεκινήσει διαδικασία επιπαραβάση ή οποιαδήποτε άλλη ενωσιακή διαδικασία όσον αφορά αυτό το θέμα. Πρέπει να σας πω ότι τέτοιου είδους ζητήματα μπορούν να ε, ε, συζητηθούν ενώπιον των εθνικών ε, δικαστηρίων που έχουν αρμοδιότητα για τέτοια θέματα. Θα προσθέσω το εξής όσον αφορά την ε, οδηγία για τα οπτικοακουστικά μέσα. Είναι γεγονός ότι εκεί περιλαμβάνονται διατάξεις οι οποίες ε, αναφέρονται στην πρόσβαση, ε, στην πληροφόρηση και την δυνατότητα, το δικαίωμα που έχουν όλοι οι ασχολούμενοι με το θέμα να μεταδίδουν τα αθλητικά γεγονότα. Αλλά στην προκείμενη περίπτωση ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να ληφθεί υπόψη το ε, ό,τι αναφέρεται στο άρθρο 15 του ιδίου κανονισμού. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, η κυρία Σακοράφα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, σήμερα έχουμε μία αναφορά που έχει σαν αντικείμενο το δικαίωμα στη διαπίστευση των εργαζομένων στα ραδιόφωνα στους αγώνες και στα αθλητικά γεγονότα. Ε, όπως ξέρουμε όλοι και όπως αναφέρθηκε οι δημοσιογράφοι είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν πολλές φορές πολύ υψηλά ε, τέλη ε, διαπίστευσης με αποτέλεσμα να έχουν δυσκολία στο να μπορέσουν να μεταδώσουν τους αγώνες. Θα μου επιτρέψετε να πω, επειδή ακριβώ υπήρξα για πάρα πολλά χρόνια αθλήτρια στο παρελθόν, όποιο ασχολείται με τον αθλητισμό γνωρίζει πάρα πολύ καλά πόσο σημαντικό είναι το ίδιο το γεγονό σαν δράση περιγραφικά μπορώ να πω να μπορεί να φτάσει στο πιο απομακρυσμένο χωριό αλλά και πόσο σημαντικό είναι ο ίδιος ο αθλητής να μπορεί να επικοινωνήσει την επικοινωνία του, την επιτυχία του και να τη μοιραστεί με όλους. Επίσης γνωρίζουμε και αναφέρθηκε προηγουμένως ότι ο αθλητισμός τα τελευταία χρόνια μια καθαρά κατά τη δική μου άποψη αραστεχνική δράση έχει γίνει ένα αντικείμενο αν θέλετε όλο και περισσότερο οικονομική συναλλαγή με αποτέλεσμα να έχουμε πολύ άσχημα φαινόμενα όσον αφορά τον αθλητισμό και να παρατηρούμε φαινόμενα τα οποία δεν συνάδουν αν θέλετε με, την αξία, με τις αξίες και το πνεύμα του αθλητισμού γενικότερα. Και αυτό γιατί παρακορήθηκε στις ομοσπονδίες και τους οργανωτές και όχι πάντα στις δημόσιες αρχές όπως αναφέρθηκε από την Επιτροπή ε, το δικαίωμα να θεσπίζουν μονομερώς τους δικούς τους κανόνες και με αυτόν τον τρόπο να έχουμε όλο και περισσότερο περιορισμούς όσον αφορά στην πρόσβαση των δημοσιογράφων, πολλές φορές των κρατικών τηλεοπτικών και ε, ραδιοφωνικών μέσων, στα αθλητικά γεγονότα, ακριβώς γιατί τα ραδιοφωνικά δικαιώματα, παραδείγματο χάρη, του Champions League όπως αναφέρθηκε, παραχωρούνται σε ομάδες που αποφασίζουν οι ίδιες σε ποιες και σε πόσους ε, ε, ραδιοφωνικούς σταθμούς θα, θα μεταδώσουν δωρεάν, ενώ τα υπόλοιπα θα πληρώσουν. Εδώ πιστεύω, κυρία Πρόεδρε, ότι υπάρχουν δύο κίνδυνοι. Ο πρώτος είναι ότι αν δεν υπάρξει άμεση παρέμβαση τώρα, το επόμενο βήμα θα είναι να ισχύσουν πραγματικά περιορισμοί στον γραπτό τρύπο και στο ίντερνετ, με αποτέλεσμα την κατάφορη καταπάτηση του δικαιώματος της ελευθερίας του λόγου και της έκφρασης της γνώμης και κατά την άποψή μου αυτό δεν συνάδει με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι το δικαίωμα της ελευθερίας της λήψης ή της μετάδοση των πληροφοριών ή των ιδεών χωρίς την ενάμειξη των δημόσιων αρχών και αδιακρίτως συνόρων συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας και της πολυφωνίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης και την πρόσβαση του Εβραίου κοινού στην ενημέρωση. Και δεύτερον, μέσα από αυτόν τον αθέμητο και ιδιόμορφο ανταγωνισμό δεν μπορεί παρά να υπάρχουν ευμενή σχόλια, δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχει κριτική σε αυτό καθ' αυτό το γεγονός. Προσωπικά πιστεύω ότι η κάλυψη των αθλητικών γεγονότων ή ακόμα και των συνεντεύξεων τύπου πριν ή μετά τους αγώνες ή οι δηλώσεις των αθλητών αν θέλετε για όσους έχουν παρακολουθήσει αγώνες στη νεκρή ζώνη, στη μεικτή ζώνη θα πρέπει να πάψουν να είναι αντικείμενο οικονομικής συναλλαγής και θα πρέπει όλοι οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι να έχουν πρόσβαση. Ε, δεν χρειάζεται να δώσω παραδείγματα γιατί τα έχουν δώσει ήδη παριστάμενοι. Απλά θα ήθελα να σας πω, γι' αυτό πιστεύω, ότι θα πρέπει η Επιτροπή να αναλάβει δράση και να γίνουν συστάσεις στα κράτη ώστε να παρεύουν σε αυτό το τόσο σοβαρό θέμα. Γι' αυτό και θα πιστεύω ότι θα πρέπει η υπόθεση να παραμείνει ανοιχτή και να την παρακολουθούμε. Σας ευχαριστώ. Thank ευχαριστώ. Ο κύριος Μαριάς. Κυρία Πρόεδρε, θεωρώ ότι η αναφορά την οποία συζητούμε είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική και έχει δύο πλευρές. Η μία πλευρά έχει σχέση βεβαίως με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα τα οποία παραβιάζονται από συγκεκριμένες ομοσπονδίες, ιδιωτικούς φορείς, επιχειρήσεις, ομάδες που έχουν σχέση και με το δικαίωμα στην ενημέρωση και με το δικαίωμα στην πληροφόρηση και με την πολυφωνία. Η δεύτερη πλευρά έχει σχέση με την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης και του άρθρου 86 την παραβίαση της συνθήκης από την πλευρά των συγκεκριμένων ομοσπονδιών. Εδώ πλέον μερικοί θεωρούν στην Ευρώπη ότι ο αθλητισμός είναι τσιφλίκι τους. Και τι συμβαίνει πρακτικά ομοσπονδίες βρίσκονται εκτός ελέγχου. Στο όνομα της δίθεν αυτοδιοίκησης των ομοσπονδιών απαγορεύεται από τα κράτη-μέλη να έχουν παρέμβαση στον τρόπο λειτουργίας αυτών των ομοσπονδιών. Κανείς και καμία νομική οντότητα δεν είναι εκτός κοινοτικού δικαίου. Οι πάντες ελέγχονται και οι συμπεριφορές και οι δραστηριότητες. Και το θέμα που θέτει η αναφορά έχει άμεση σχέση και με οικονομικά δικαιώματα. Διότι οι συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι ασκούν μια οικονομική λειτουργία. Και η οικονομική λειτουργία την οποία ασκούν προστατεύεται από τις διατάξεις της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι το δικαίωμά τους και ως εργαζόμενοι να ενεργούν ελεύθερα και ως πάροχοι υπηρεσιών και ταυτόχρονα δεν πρέπει να υπάρχουν ομοσπονδίες οργανισμοί οι οποίοι καταχρώνται τη δεσπόζουσα θέση την οποία έχουν αυτή τη στιγμή. Ήρθε η ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει μία μεγάλη έρευνα και απευθύνομαι στην Κομισιόν, στη Διεύθυνση Ανταγωνισμού. Θα πρέπει να ελεγχθεί αν η FIFA, η UEFA, οι διάφορες ομοσπονδίες ποδοσφαίρου και αθλητισμού ενεργούν καταχρώμενες τη δεσπόζουσα θέση την οποία έχουν. Βγάζουν αποφάσεις οι οποίες δεν ισχύουν μόνο ως κανονισμοί λειτουργίας σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις όπως είναι το Champions League, αλλά οι αποφάσεις τους ισχύουν και για τη λειτουργία των πρωταθλημάτων σε κάθε κράτος μέλος. Και έχουμε λοιπόν παρέμβαση με τρόπο που στόχο έχει τον περιορισμό του ανταγωνισμού τον περιορισμό της δυνατότητας ποδοσφαιριστών ή άλλων αθλητών να μεταγράφονται ελεύθερα. Και όλα αυτά γίνεται για να προστατευτούν πολυεθνικές ποδοσφαιρικές ομάδες ή ομοσπονδίες τα έσοδά τους. Ήρθε λοιπόν η ώρα και το λέω ότι πρέπει να αναλάβουμε ίσως και εμείς εδώ ως Επιτροπή μια πρωτοβουλία. Να σταματήσει αυτή η ιστορία. Δεν μπορεί να είναι έξω από τον έλεγχο του νόμου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών αυτές οι ομοσπονδίες. Διότι έχει δημιουργηθεί μια γκρίζα ζώνη, μια γκρίζα ζώνη μη ελέγχου, η οποία έχει αυτά τα αποτελέσματα που είδαμε. Να απαιτούν τεράστια ποσά για τη διαπίστευση. Άρα λοιπόν να παραμείνει ανοιχτή η υπόθεση αυτή και πιστεύω ότι η επιτροπή πρέπει να είναι πιο αποφασιστική απέναντι σε αυτές τις λειτουργίες των ομοσπονδιών που καταχρώνται τη δεσπόζουσα θέση τους στην ευρωπαϊκή ένωση. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ζητήσω από όλους τους συναδέλφους να είναι λίγο πιο σύντομοι από ό,τι είσαστε εσείς κυρία Μαριά, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Η κυρία Λίτιγκερ. Λίδια, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν θα επαναλάβω όσα υπόθηκαν ήδη. Έχω μεγάλη εμπειρία επί του θέματος ε, γιατί ήμουν δημοσιογράφος ε, και μάλιστα διευθύντρια στην πολωνική τηλεόραση. Επομένως γνωρίζω πάρα πολύ καλά το πρόβλημα το οποίο συζητάμε σήμερα. Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι δυνατόν μέσω ατραπών να ξεφεύγει από τις ευθύνες της. Δεν είναι δυνατόν να λέει ότι δεν εντάσσεται στις αρμοδιότητές της το ζήτημα αυτό, μια και πρόκειται για το δικαίωμα που έχει κάθε ένας Ευρωπαίος πολίτης για πρόσβαση στην ε, πληροφορία. Ε, επομένως, μέσω των δημοσιογράφων πρέπει να περνάει η πληροφόρηση στους Ευρωπαίους πελίτες. Έχουμε ακούσει εδώ ότι, ας πούμε, στη Γαλλία η κατάσταση είναι διαφορετική, ενώ ε, γνωρίζουμε ότι σε άλλες χώρες, πέρα από τη Γαλλία, η διαπίστευση κοστίζει πάρα πολύ ακριβά στους δημοσιογράφους. Οπωσδήποτε θα πρέπει να γίνει κάτι φυσικά. Ε, στην ε, Ευρώπη έχουμε πάρα πολλούς οι οποίοι ασχολούνται με το θέμα αλλά στον ε, ιδιωτικό τομέα. Ωστόσο θα πρέπει να υπάρξει μια ρύθμιση από πλευράς της Επιτροπής. Κυρίως όσον αφορά όπως είπαμε την διαπίστευση θα πρέπει να ακολουθήσουμε ενδεχομένως το δρόμο που είχαμε ακολουθήσει για το θέμα της περιαγωγής, για το θέμα των κινητών τηλεφώνων και της χρέωσης των συνδιαλέξεων. Νομίζω ότι και εδώ θα πρέπει να αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει κάτι αντίστοιχο. Όπως τα κινητά βάλαμε ε, ένα, ε, μια συγκεκριμένη ε, χρέωση, θα πρέπει να υπάρχει μια αντίστοιχη δυνατότητα ενιαίας χρέωσης και στην πληροφόρηση. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Μαρτά. Παρακαλώ κύριε Μαρτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η απάντηση της Κομισιόν δεν με εκπλήσει. Μάλιστα πρέπει να πω δεν με εκπλήσει καθόλου. Γιατί σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι η Ευρώπη θα πρέπει να είναι μια μεγάλη αγορά και επομένως το μόνο ζήτημα που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της απαντήσεώς της είναι εάν ε, και η πληροφόρηση είναι όχι απλώς ένα ε, εμπόρευμα, αλλά ένα εμπόρευμα του χειρίστου είδους. Και από την άλλη πλευρά θα πρέπει να δούμε αν και κατά πόσον ισχύει η, ισονομία μεταξύ και η ισότητα μεταξύ των πολιτών. Ε, γιατί αυτή τη στιγμή ε, το, η μετάδοση των αθλητικών διοργανώσεων είναι το μόνο που έχει απομείνει στους πιο φτωχούς πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι δυνατόν να πληρώνουμε λοιπόν εκατομμύρια, ε, δεκάδες, εκατοντάδες εκατομμύρια ε, για τα, ε, για τα δικαιώματα αυτά και εν τέλει να καταλήγουμε οι Ευρωπαίοι πολίτες ή τέλος πάντων η μεγάλη πλειοψηφία των Ευρωπαίων πολιτών να μην έχει πρόσβαση σε αυτά τα αθλητικά γεγονότα γιατί οι διοργανώσεις αυτές θα γίνονται πλέον πάρα πολύ ακριβές. Νομίζω ότι σαν Ευρωπαίοι βουλευτές και εμείς οφείλουμε να ξεκινήσουμε ξεκινήσουμε μια λαϊκή διαβούλευση, μια λαϊκή διαδικασία έτσι ώστε να απαιτήσουμε κάποια πράγματα και να απαιτήσουμε βεβαίως ε, και το fair play γιατί αυτό το fair play έχει γίνει καραμέλα στο στόμα όλων των υψηλά ισταμένων αθλητικών παραγόντων. Να γίνει ουσία τουλάχιστον. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα και εγώ. Σαφώς εδώ μας λέει η Επιτροπή ότι δεν είμαστε αρμόδιοι. Εμάς δεν μας ικανοποιεί αυτή η απάντηση, δεν μας ικανοποιούν αυτά που συμβαίνουν και εμείς λέμε όχι. Το θέμα είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν μας δόθηκαν οι πληροφορίες που ζητήσαμε και αυτό που θέλουμε είναι να σταλούν αυτά τα στοιχεία στις αρμόδιες επιτροπές. Είναι θέμα εσωτερικής αγοράς, θέμα δίκαιου ανταγωνισμού, δεν ξέρω ακριβώς, αλλά σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε το δικαίωμα για έμεση αναφορά. Πρέπει να αλλάξει κάτι εδώ και ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει κάποιες ε, αποφάσεις ε, νομοθετικές, κανονιστικές. Ε, εμείς, αν αυτό δεν γίνει, θα απευθυνθούμε στις αρμόδιες επιτροπές. Θα δούμε με τους άλλους συναδέλφους ποιες είναι οι υπόλοιπες κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες τις οποίες μπορούμε να αναλάβουμε αν δεν είναι ικανοποιητική η δράση της Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Νομίζω ότι αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε θα δώσω βέβαια το λόγο πάλι στους αναφέροντες. Πολύ σύντομα όμως, σας παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, ειδικά τους Ευρωβουλευτές, επειδή πιστεύω ότι κατανόησαν το πρόβλημα το οποίο εστιάζεται στο δικαίωμα της πληροφόρησης των φτωχών Ευρωπαίων πολιτών, της άμεσης πρόσβασης με τους αθλητές. Οι αθλητές είναι το νόημα του αθλητισμού και με την επιβολή τελών ή απαγορεύσεων στις μειχτές ζώνες και στη συνέντευξη τύπου μας αποκλείουν την πρόσβαση με τους αθλητές, αποκλείουν την επικοινωνία του Ευρωπαίου πολίτη με τον πρωταγωνιστή που είναι αθλητής. Είμαστε εξαιρετικά απογοητευμένοι από την θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν είναι όλα εμπόρευμα δεν είναι όλα προς αγορά και πώληση. Υπάρχουν και δικαιώματα για τους αθλητές, για τους δημοσιογράφους, για τους Ευρωπαίους πολίτες. Και πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σας ευχαριστούμε σαν Ευρωβουλευτές να πάρετε πρωτοβουλίες. Δεν είναι όλα εμπορεύματα. Δεν είναι όλα να έχουμε έναν πάγκο έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τα αγοράζουμε και να τα πουλάμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. So, my proposal would be... Η πρότασή μου είναι, βεβαίως, όπως είπε η κυρία Σακοράφα, ο Πίτερ Γιάρ και άλλοι, παραμένει ανοιχτή η αναφορά σας και μπορούμε, μπορούμε, και ίσως αυτό είναι και το καλύτερο, να απευθυνθούμε στην αρμόδια επιτροπή που είναι η Επιτροπή Πολιτισμού και Αθλητισμού να τους ζητήσουμε να γνωμοδοτήσουν βάσει της δικής τους γνωμοδότησης θα ακολουθήσουμε την ορθότερη οδό. Αυτή τη στιγμή υπάρχει δυνατότητα, το προβλέπει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, να κάνουμε κάτι Ακριβώς επειδή κάτι δεν υπάρχει στην οδηγία για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εμείς μπορούμε παρόλα αυτά να το λάβουμε υπόψη μας. Αυτή είναι λοιπόν η πρότασή μου. Συμφωνείτε όλοι? Μπορεί επίσης να σταλεί στην Επιτροπή ε, αναφορά και στην Επιτροπή που είναι αρμόδια για τα θέματα ανταγωνισμού και εσωτερικής αγοράς επίσης. Okay. Εντάξει, εντάξει, ωραία και στην Επιτροπή Πολιτισμού και Αθλητισμού και στην Επιτροπή εσωτερική αγορά και Ανταγωνισμού. Βάσει των γνωμοδοτήσεων αυτών των δύο επιτροπών θα πάρουμε την απόφασή μα για τη συνέχεια, είτε έκθεση πρωτοβουλία, αλλά κάτι θα κάνουμε. Σίγουρα όμω, Ήθελα να σας πω, ευθύνομαι στους αναφέροντες, ότι θα ασχοληθούμε με το θέμα σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σας ευχαριστώ πολύ. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι τώρα το 8. Πρόκειται για την έκθεση του Λούις Χάρτ 1569 και μια σειρά άλλων αναφορών. Δεν θα δώσω τώρα ε, τις τίτλους όλων αυτών των αναφορών. Υπάρχουν στην ημερήσια διάταξη. Η Ρελά Τελέλη από την Ιταλία είναι εδώ. Πού είναι? Εδώ είστε. Καλωσορίσατε. Η Επιτροπή είναι επίσης εδώ. Επίσης, και το Συμβούλιο. Ωραία, περνάμε λοιπόν τώρα σε ένα τελείως διαφορετικό θέμα. Θέλω να πω στους προηγούμενους αναφέροντες, μπορείτε αν θέλετε να μείνετε ή να εγκαταλείψετε την αίθουσα. Το θέμα σας ε, το εξαντλήσαμε. Και τώρα περνάμε σε θέματα μετανάστευσης. Ρενάτο Λέλη είναι ο πρώτος που θα πάρει το λόγο. Καλή σας μέρα πρόεδρος της Ένωσης Διαζευμένων Γονέων ε, από την Βερόνα. Κυρία Πρόεδρε, κύριοι βουλευτές, θα είμαι σαφής. Εμείς οι Ευρωπαίοι πολίτες ε, και οι πολίτες της Ιταλίας ε, προβληματιζόμαστε ιδιαίτερα. Όλοι υψώνουν όλες οι χώρες ε, ε, υψώνουν ε, τα τείχη τους έτσι ώστε να εμποδίσουν την μετανάστευση εκτός από την, την Ιταλική κυβέρνηση, τη μία εκλεγμένη η οποία επιτρέπει σε όλους να περάσουν τα σύνορα. Με έναν τεράστιο αριθμό ανέργων παρόλα αυτά η χώρα μου επιτρέπει αδιακρίτως την μεταναστευτική ε, που δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Γι' αυτό λοιπόν εμείς ζητούμε με ταχύτητα ε, να ληφθούν αποφάσεις έτσι ώστε να σταματήσει άμεσα η επιχείρηση Mare Nostrum. η κατάσταση. Από τον Οκτώβριο του 2013 μέχρι τώρα στην Ιταλία έχουμε υποδεχθεί 130 λαθρέους παράνομους μετανάστες. Ε, τα χρήματα τα οποία έχουν δοθεί ανέρχονται σε πολλά εκατομμύρια που θα μπορούσαν να είχαν χρησιμοποιηθεί ε, έτσι ώστε να βοηθηθούν οι φτωχοί, οι άποροι, οι αποκλεισμένοι και οι άνεργοι της χώρας μου ε, που ε, εν πάση περιπτώσει θα μπορούσαν ε, να χρησιμοποιηθούν έτσι ώστε να ανεβεί λίγο το ΑΕΠ μας και το ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ήθελα να πω ότι το πρόβλημα αυτό δεν είναι μόνο ιταλικό, είναι πρόβλημα ενωσιακό, είναι πρόβλημα παγκόσμιο. Αυτή η επιχείρηση του Μάρε που οργανώθηκε από τον προηγούμενο ε, πρωθυπουργό ε, Μάριο Λέτα ενδίκολετα Λέτα, ε, είναι μια επιχείρηση η οποία είναι και στρατιωτική και πολιτική και η οποία υποτίθεται ότι ελήφθη εν αναμονή κάποιας άλλης ε, απόφασης και κάποιας άλλης επιχείρησης. Ωστόσο, οι ε, πόλεμοι στην Συρία, η επικίνδυνη κατάσταση στην Αίγυπτο, στην Συρία, στην Τουρκία αποτελούν πολύ μεγάλη απειλή πλέον. Απειλείται η Ήπειρός μας, διότι μέσω αυτών των ε, ε, ροών ε, ξανά θυμόμαστε αρρώστιες ξεχασμένες όπως η φυματίωση, η ελονοσία κλπ. Για να μην πω για το έμπολα που αρχίζει τώρα και χτυπάει τις πόρτες μας. Ακόμα και ε, χτες ε, ε, πιάσανε η Guardia di Finanza πλοία μεταναστών γεμάτα λαθρέα εμπορεύματα και ναρκωτικά. Έχει τριπλασιαστεί το, το, ο αριθμός των ναρκωτικών που, βρίσκονται, που έχουν κατασχεθεί από την Guardia di Finanza. Δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε πλέον την κατάσταση αυτή. Δεν είναι δυνατόν λόγω του υψηλού μας χρέους να δεχτούμε τέτοιου είδους, τέτοιου είδους ε, ε, καταστάσεις. 20 δευτερόλεπτα δεν είναι δυνατόν να δώσουμε τα έξοδα αυτά. 10 ε, εκατομμύρια τον ε, μήνα δίνονται για την ε, βοήθεια αυτών των ανθρώπων, ενώ τα χρειάζεται η Ιταλία. Δεν είναι δυνατόν επίσης να δεχτούμε την πλήρη αποτυχία του Μάρε Νόστρουμ, η οποία έχει επιστεγαστεί από τόσους θανάτους. Λοιπόν, θεωρούμε ότι θα πρέπει να δώσουμε μονάχα σε κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις τα δικαιώματα δικαίωμα ασύλου μετά από πάρα πολύ μεγάλο έλεγχο. Επίσης, 18 Οκτωβρίου στο ε, Μιλάνο θα οργανωθεί μια μεγάλη διαδήλωση για να σταματήσει αυτή η ανεξέλεγκτη και λαθρέα μετανάστευση. Να σα σχολιάσω, very... να σας σχολιάσω σύντομα ότι εδώ στο σώμα μας αυτό είναι σημαντικό να πούμε ότι κανένας ε, άνθρωπος, κανένα ανθρώπινο όν δεν είναι παράνομο. Έτσι, αυτό θα ήθελα να το τονίσω. Και αυτό νομίζω ότι αφορά τη θέση όλου του Κοινοβουλίου. the Τώρα με χαρά να δώσω το λόγο στον Φιλίπ Κολόμπο ή στον Τζενάρο Κάπο από την Ιταλική Μονιμή Αντιπροσωπεία. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Είμαι ο Φίλιππο Κολόμπο από τη μόνιμη Ιταλική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαι εδώ λόγω της Ιταλικής Προεδρίας. Τα ερωτήματα που θέτει ο Δόκτωρ Λέλη αφορούν μία από τις προτεραιότητες της Προεδρίας μας. Θα έχουμε το Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων σε λίγες ημέρες στο Λουξεμβούργο. Οι Υπουργοί Εσωτερικών θα συναντηθούν την Πέμπτη και στην ημερήσια διάταξη υπάρχει το θέμα των μεταναστευτικών ροών, ιδιαίτερα της μεταναστευτικής πίεσης. Ιδιαίτερα βέβαια όσον αφορά την κεντρική Μεσόγειο. Η Ιταλική Προεδρία, σε συμφωνία με την Κομισιόν και τις χώρες μέλη, πρότεινε μια νέα προσέγγιση με τρεις πυλώνες που συζητήθηκε στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ ξεκίνησε ένα βίντεο δυστυχώς ταυτόχρονα. We apologize for that. Ζητώ συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη, παρακαλώ, συνεχίστε. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Έλεγα λοιπόν ότι έχουμε μια προσέγγιση με τρεις πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας αφορά την δράση σε συνεργασία με τις χώρες μέλη. Ο δεύτερος πυλώνας αφορά την ενίσχυση του Frontex και των δράσεων επιτήρησης και ελέγχου των συνόρων και ο τρίτος πυλώνας αφορά την υποδοχή, το fingerprinting που λέμε, δηλαδή την καταγραφή των ατόμων όταν φτάνουν στην Ευρώπη. κύριος Λέλη αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο Μάρε Νόστρομ να του πω ότι όπως είπε και ο κύριος Λέλη, το Μάριο Νοροστρούμ αφορά μια έκτακτη κατάσταση και έτσι το βλέπουμε εμείς. Εμείς θα θέλαμε και ως προεδρίες αυτό εργαζόμαστε να ξεπεραστεί αυτή η κατάσταση έκτακτης ανάγκης και να υπάρχει μια προσέγγιση πιο βιώσιμη όσον αφορά την διαχείριση της μεταναστευτικής πίεσης. Για την Κεντρική Μεσόγειο Καθορίζουμε τώρα τις νέες δράσεις Frontex που ελπίζουμε να οδηγήσουν στην υπέρβαση, στο να ξεπεραστεί δηλαδή η επιχείρηση Mare Nostrum. Για την Ιταλική λοιπόν Προεδρία, προς το παρόν, αυτές είναι οι προτεραιότητες μας. Και βεβαίω είμαστε στη διαθεσή σας για περαιτέρω διευκρινήσεις και για τους ε, κύριους ευρωβουλευτές αλλά και για τον ε, Ετώντα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κολόμπο. Μιλήσατε εξ ονόματος της Ιταλικής αντιπροσωπείας, μόνης αντιπροσωπείας, ο Τζενάρο Κάπο, ένα άλλο όνομα έχω εγώ. Ναι, ναι, είναι συνάδελφος, αλλά ναι, μιλήσατε εξ ονόματος και των δύο. Χαίρομαι. Ωραία. Ο κ. Ματίας Ερλ έχει το λόγο μέσα στις Κομισιόν. Thank you very much, uh, Madam Πρόεδρε, ευχαριστώ. Το θέμα που έχουμε σήμερα περιλαμβάνει εννέα αναφορές που ασχολούνται με το ίδιο ζήτημα, την αποτροπή τραγωδιών όπως αυτές που έγιναν πέρσι, όπως αυτή που έγινε πέρσι στη Λαμπεντούζα. Οι πληροφορίε που έδωσε η Κομισιόν αφορούσαν την περσινή τραγωδία, οπότε με χαρά να ενημερώσω την Επιτροπή σας για το τι έχει μεσολαβήσει. Και αφού η αναφορά αφορά κυρίως τη Μεσόγειο, να σας δώσω έτσι μια σύντομη επισκόπηση για τη δουλειά που κάνει αυτή η Task Force. Η Task Force για τη Μεσόγειο συγκροτήθηκε από το Συμβούλιο του Οκτώβρη, αμέσως μετά δηλαδή την τραγωδία στη Λαπεντούζα, λίγες μέρες μετά και αποτελείται από την Κομισιόν, χώρες μέλη, κοινοβούλιο, οργανισμούς με κυβερνητικού κλπ. Και στόχος της Επιτροπής αυτή ήταν το να εντοπίσει βάσει ακριβώς των αρχών της πρόληψης, της ελεγγύης κλπ δράση προτεραιότητα, για να γίνουν πιο αποτελεσματικά τα εργαλεία και οι πολιτικές της Ένωσης ώστε να αποτραπεί το ενδεχόμενο τέτοιων τραγωδιών στο μέλλον. Τώρα ποια είναι η πολιτική πρόκληση, οι προκλήσει, πρόεδρε. Είναι το να μην κάνουν ταξίδια ρηψοκίνδυνα, επικίνδυνα για τη ζωή τους οι μετανάστες στη Μεσόγειο. Δηλαδή να μην μπαίνουν με σκάφη από τις βόρειες ακτές της Αφρικής το οποίο σημαίνει ότι οι περισσότερες δράσεις που θα πρέπει να αναλάβουμε πρέπει να λάβουν χώρα σε συνεργασία με τις χώρες μετακόμισης και με τις χώρες προέλευσης στην Αφρική. Η Task Force για τη Μεσόγειο αποτελεί ένα παράδειγμα κατά την άποψή μου το πώς η Ευρώπη μπορεί να αντιδράσει. Γιατί έξι μέρες αργότερα μετά τη σύστασή της συνέταξε μια πολύ επτομερή έκθεση όπου εντοπίστηκαν διάφοροι τομείς δράσης και υποβλήθηκαν στην Ιταλική Προεδρία. Οι δράσεις που έχουν αναλυφθεί από το Συμβούλιο και την ε, Προεδρία είναι πλήρως ευθυγραμμισμένες με τη δουλειά της Task Force. Να σας ενημερώσω τουλάχιστον για τις πέντε αυτές περιοχές οι οποίες είναι σύμφωνες με αυτούς τους στόχους, δηλαδή συνεχίσαμε με τις χώρες, ενίσχυση του προγράμματος παρακολούθησης, καταπολέμηση ε, του λατρεμπορίου, επιτήρηση των συνόρων και αρρωγή και αλληλεγγύη με άλλες χώρες μέλη. Θα ήθελα να σας δώσω κάποια παραδείγματα για το τι έχει πετύχει η Task Force αυτή μέχρι τώρα στο διάστημα που μεσολάβησε το έτος βάσει των, της έκθεσης της Task Force. Πολλές από τις δράσεις ήδη έχουν αναπτυχθεί και ή βρίσκονται στην φάση εφαρμογής η πρόοδος να ήταν αργή, είναι όμως σταθερή και σχετίζεται ευρέως με το γεγονός ότι εμείς συζητάμε για... και μιλάμε με δύσκολες κυβερνήσεις, Λιβύη, Αίγυπτος, όπου είναι δύσκολο να επιτευχθεί ταχεία πρόοδος. Θετικές εξελίξεις είχαμε πάντως. Να σας δώσω παράδειγμα σύντομα. Ένας διάλογος πολιτικής με την Ανατολική Αφρική έχει ξεκινήσει και είχαμε στο Χαρτούμ υπουργική συνάντηση. Θα έχουμε τον Οκτώβριο, τέλειο Οκτώβριο και Νοέμβρη στη Ρώμη. Έχουμε επίσης και συμφωνία με την Ιγυρία. Έχουμε επίσης ε, συμφωνίες κινητικότητας με το Μαρόκο και την, την Ισία που, θα έχουν, που έχουν εφαρμοστεί και θα υπάρξουν και άλλες συμφωνίες για να υποστηρίξουμε το Μαρόκο όσον αφορά τα θέματα ασύλου. Είχαμε μια, σχέση εταιρικής, μια συμφωνία εταιρική σχέση με την Ιορδανία που επικυρώθηκε από το Συμβούλιο. Μάλλον που θα επικυρωθεί από το Συμβούλιο αυτή την εβδομάδα. Έχουμε επίσης και με το Λίβανο διάλογο, κάτι το οποίο συζητείται και με τις χώρες μέλη. Τώρα τα προγράμματα προστασίας για το κέντρο Αφρικής και τη Βόρεια Αφρική είχαν συζητηθεί πρόσφατα μόνο με τις χώρες μέλη. Πρόθεσή μας είναι να ενισχύσουμε αυτά τα προγράμματα περιφερειακής προστασίας και να επεκταθούν σε όλη την Βόρεια Αφρική, συμπεριλαμβανομένων και διάφορων δράσεων με την συμμετοχή των χωρών μελών. Οι εκστρατείες μας θα ξεκινήσουν βεβαίως στις κύριες χώρες διαμετακόμισης, στην μεταναστευτική οδό στην Ανατολική και Δυτική Αφρική σε συνεργασία με τον ΟΙΕ. Άλλη ως ένας τομέας προτεραιότητας είναι η ανάπτυξη σχεδίου συνεργασίας για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου σε σχέση και συνεργασία βέβαια με τις χώρες της περιοχής ιδιαίτερα αυτές με διαμετακόμισης και τέλος για την ανθρωπιστική υποδοχή. Αυτό παραμένει προς το παρόν ο κύριος τρόπος προστασίας μας για τα άτομα που εισέρχονται στην Ένωση για την νομική τους προστασία. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε τύχη Θέλουμε να υπάρχουν νόμιμες είσοδοι, οδές, συγγνώμη, εισόδου στην Ευρώπη. Θα ήθελα τώρα να περάσω στο θέμα των συνόρων. Όπως είπε και ο αναφερόμενος, έχουμε την δράση Mare η οποία έχει καθαρά εθνικό χαρακτήρα και πρόσφατα είχαμε μια προκατακτική συμφωνία μεταξύ Ιταλίας και Frontex για την ενίσχυση ε, Τη Τρίενα, της επιχείρηση Τρίενα που θα ξεκινήσει τον Νοέμβρη. Ελπίζω η σύντομη αυτή επισκόπηση που σας έκανα να σας δείχνει σωστά την προσέγγισή μας για την αποτροπή των τραγωδιών αυτών στην ε, Ευρώπη με ολοκληρωμένο τρόπο ώστε να παραλαμβάνονται και εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές και πολιτικές συνεργασίες και συνεργασία με άλλους εμπλεκόμενους ε, μη κοινωνικέ οργανώσεις κτλ. Θα πρέπει λοιπόν να αποφύγουμε την ε, διεξαγωγή ταξιδίων με θάνατο, με κίνδυνο για τη ζωή τους από τους μετανάστες, δουλεύοντας και με τις χώρες μετακόμισης και με τις χώρες προέλευσης. Η πρόοδος δεν είναι εύκολη, αλλά ελπίζω η επισκόπηση αυτή να σας έδειξε ότι είναι σταθερή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ γιατί πραγματικά μας περιγράψατε ποιες είναι οι προκλήσεις που έχουμε απάντησή μας καθώς και το θέμα των ασφαλών οδών για, αυτόν τον, για αυτούς τους πρόσφυγες, για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να εγκαταλείψουν τις πατρίδες τους. Σαφώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθούμε να πετύχουμε κάτι. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για το πραγματικά ευρωπαϊκό σας πνεύμα. Ο τρόπος που αντιμετωπίζετε αυτό το θέμα είναι πραγματικά ευρωπαϊκός. Και θα ήθελα εδώ να αναγνωρίσω πραγματικά τις αρχές της Ιταλίας, οι οποίες έχουν σώσει χιλιάδες, χιλιάδες ζωές με το Mare με τη γενοδορία τους, με την ανθρωπιστική προσέγγιση. Είναι δύσκολη η κατάσταση και όλοι ξέρουν ότι πάνω από 18.000 ζωές συγγνώμη, 80.000 ζωές ή 100.000 ζωές έχουν σωθεί από τους Ιταλούς, από τις αντιλικές αρχές. Και πρέπει να το αναγνωρίσουμε και να μιλήσουμε για την γενεοδορία του Ιταλικού λαού. Υπάρχουν βέβαια διαφορετικές απόψεις για το θέμα αυτό, αλλά αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι εμείς σαν Επιτροπή Αναφορών δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να βρεθούμε σε μια μεροληπτική στάση. Η στάση μας είναι σαφής. Ο καθένας μπορεί να βλέπει κάπως διαφορετικά το θέμα της μετανάστευσης, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει εδώ είναι να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας την κάθε αναφορά. Να προστατέψουμε δηλαδή το δικαίωμα να υποβάλλονται αναφορές όλους. Και τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε την συζήτηση. Η κυρία Τζοφρίντα έχει ζητήσει το λόγο. Ε, Ευχαριστώ. Αναφέρομαι, θα αναφερθώ μάλλον σε αυτά που μόλις είπατε, γιατί σημαίζομαι απόλυτο όχι μόνο το πνεύμα, αλλά και την προσέγγιση για αυτό το είδος προβλήματος. Εμείς δεχτήκαμε δεκάδες ερωτήματα από τους πολίτες μας, Ευρωπαίους πολίτες που πραγματικά ανησυχούν πολύ. Στο συγγνώμη που απουσίαζα πριν από λίγο και δεν άκουσα την ε, προηγούμενη εισαγωγική παρέμβαση. Είναι όμως σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι η προσέγγιση, τουλάχιστον η προσέγγιση, πρέπει να είναι κοινή όσον αφορά αυτή την ανθρωπιστική τραγωδία. Δεν έχουμε να κάνουμε με ένα θέμα διαμάχης μεταξύ χωρών. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε λάβει και τόσες αναφορές για αυτό το θέμα, όπως υπόθηκε προηγουμένως. Πολλές από αυτές τις αναφορές αναφέρονται στην φάση μετά από αυτή την τραγωδία Λαπεντούζα, που έγινε πριν ένα χρόνο. Και σε σχέση με αυτή την τραγωδία ακολούθησαν εκατοντάδες άλλων θυμάτων, το οποίο σημαίνει ότι δεν καταφέραμε να βρούμε μια λύση να βρούμε μια λύση θα ήταν κάτι το φιλόδοξο, γιατί είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι δύσκολο να λυθεί. Οπότε θα πρέπει να βρούμε μια κοινή και συγκεκριμένη προσέγγιση στο πρόβλημα αυτό. Και κυρίως θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να καταλάβουμε την διάσταση του προβλήματος. Πριν από λίγο άκουσα να γίνεται λόγος για την Task Force για την Μεσόγειο. Θα ήθελα να μάθω το περιεχόμενο της έκθεσης του εγγράφου που αναφέρθηκε και κυρίως τα αποτελέσματα της δουλειάς που έγινε. Νομίζω είναι σημαντικό στην Επιτροπή Αναφορών μαζί με τους αδέλφους της ΛΥΜΠΕ να τα γνωρίζουμε όλα αυτά. Εμείς λοιπόν πρέπει να είμαστε σε θέση να τα γνωρίζουμε όλα αυτά ακριβώς για να απαντήσουμε στους πολίτες που απευθύνονται σε εμά. Οι πρόσφατες αντιδράσεις σε σχέση με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου Σούλτς και την είπατε εκπρόσωπο Μογκερίνη δείχνουν ότι το κλίμα που αφορά που δημιουργήθηκε μετά την Λαμπετούζα είναι όλο και πιο θερμό ιδιαίτερα στην Νότια Ιταλία. Ο πληθυσμό έχει φτάσει στα ωριά του γιατί ο πληθυσμός ιδιαίτερα της Νότιας Ιταλίας βαραίνεται ή τον βαρύνει ένα πρόβλημα από ένα πρόβλημα το οποίο τονίζω είναι όλο και πιο ευρωπαϊκό, δεν είναι μόνο ιταλικό. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο ζητάω να αναλυφθεί ευρύτερα το πρόβλημα αυτό. Και είπαμε στην κυρία Μάλστρομ την Επίτροπο να υπάρξει αύξηση των κονδυλίων της Frontex, αλλά να υπάρχει αύξηση της προσοχής που θα δοθεί σε αυτό το θέμα αυτό και να υπάρχει μια αποκεντρωμένη έδρα ελέγχου εκτάκτων καταστάσεων στη Σικελία. Έγινε λόγος για το μάρενόστρουμ Nostrum και την προσεχή επιχείρηση Τρίανα. Θα αποτιμήσουμε τα αποτελέσματα γιατί όπως υπενθύμησε και ο εκπρόσωπος της κυβέρνησής μας έχουμε να κάνουμε με ενίσχυση των περιπολιών. Πρέπει όμως ταυτόχρονα να δώσουμε και απαντήσεις στα ερωτήματα του πληθυσμού που μόνος το αντιμετωπίζει το φαινόμενο αυτό στην ουσία. Κάτι το οποίο οδηγεί σε ρατσιστικές αντιδράσεις. Γι' αυτό πρέπει να κατανοήσουμε και την αντίδραση του πληθυσμού αλλά και τον αντίκτυπο που θα μπορούσε να έχει αυτό το θέμα και σε θέματα δημόσιας τάξης. Εμείς λοιπόν θα πρέπει να αντιδράσουμε και ζητώ από τους συναδέλφους να τοποθετηθούν σε σχέση με αυτό γιατί αποτελεί ένα τεράστιο πρόβλημα. Μιλάμε για μια τραγωδία την οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε δίνοντας συγκεκριμένα απαντήματα σε αυτούς που απευθύνονται σε εμά ως Επιτροπή. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Ο Grazie, Presidente. Intanto... Πρόεδρε, ευχαριστώ. να συγχαρώ την Επιτροπή για αυτή την ανοιχτή και ειλικρινή συζήτηση. Σημαντικό νομίζω είναι να ακουστεί η φωνή των πολιτών αλλά και να προσεγγίσουμε το πρόβλημα αυτό χωρίς παροπίδες ιδεολογικές. Η αναφορά του δόκτρος Λέλλη νομίζω ότι ανοίγει πραγματικά ένα σημαντικό έτσι, παράθυρο Όταν δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει σημαντικές απειλές σε σχέση με την τρομοκρατία και την εσωτερική ασφάλεια. Εγώ νομίζω ότι πέρα από τα τυπικά θέματα όπως είπε σωστά προσφόρηση της Κομισιόν εμείς πρέπει να δημιουργήσουμε ασφαλείς οδούς μετανάστευσης το οποίο σημαίνει ότι σήμερα πάρα πολλέ οδοί μετανάστευση είναι παράνομες. Θεωρώ ότι το πραγματικό πρόβλημα, οι προβλήματα είναι πραγματικά δύο. Τα οποία αφορούν ακριβώς το σωστό αίτημα για την διακοπή της επιχείρησης Μάρε Καταρχά το θέμα της ασφάλειας. Γιατί αυτό το είπαν και οι ευρωπαϊκές αρχές. Ότι δηλαδή από τις 130.000 πρόσφυγες ή άτομα τέλος πάντων τα οποία φτάνουν στο νότο της χώρας μας μόνο ένα μικρό τμήμα εντοπίζεται. Αυτό απορρέει από επίσημες δηλώσεις και όλα αυτά σχετίζονται με το συναγερμό που σήμανε ο ίδιος ο Επίτροπος για θέματα ασφαλείας στην Ευρώπη, δηλαδή 3.000 πολεμιστές του Αλάχ, τσιχαντιστές που ετοιμάζονται να μπουν στην Ευρώπη. και οι οποίοι από ό,τι φαίνεται μπορούν να ακολουθήσουν αυτές τις παράνομες οδούς μετανάστευσης. Το δεύτερο πρόβλημα που υποβόσκει στην ε, αναφορά είναι το θέμα της ασφάλειας που αφορά την αποβίβαση ατόμων ασθενών, πιθανώς δηλαδή επικίνδυνων. Ξέρετε ότι η Λαμπεντούζα δεν έχει καν νοσοκομείο, οπότε να μην κάνουμε την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη να πιστεύει ότι ελέγχονται αποτελεσματικά αυτοί οι μετανάστες για ασθένειες όπως έμπολα. Αυτό δεν ισχύει στην μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων, ιδιαίτερα σε αυτή την κατάσταση έκτακτη ανάγκη. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι είναι ε, πολύ σωστό το αίτημα για πάυση της επιχείρησης Mare Nostrum, ε, διότι ούτως ή άλλως δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Μποργέζα. Νίλ Σεμπάγιας, ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι είναι πάρα πολύ θετικό το ότι συζητούμε αυτό το θέμα. Γιατί βεβαίω είναι ένα θέμα που αφορά και το πολιτικό επίπεδο αλλά και τους πολίτες. Πολλοί αντιμετωπίζουν αυτό το θέμα σαν κάτι που αφορά όλους μας. Υπάρχουν πολλοί αριθμοί αυξανόμενη αριθμή όσον αφορά τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Πολλοί αναγκάζονται να φτάσουν στην Ευρώπη, όχι επειδή το επιλέγουν, αλλά επειδή δεν έχουν άλλη δυνατότητα, δεν μπορούν να ζήσουν στις χώρες τους. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε να τους υποδεχτούμε αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται παραδείγματος χάρη από το Ιράκ ή από τη Συρία έρχονται να βρουν καταφύγιο οι άνθρωποι αυτοί στην Ευρώπη και σαφώς και έχουμε ευθύνη που απορρέει από το διεθνές δίκαιο να προσφέρουμε άσυλο στους ανθρώπους αυτούς. Θα πρέπει επίσης να κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε να υπάρξει ειρήνη στην Συρία και στο Ιράκ και να μην υπάρχει πλέον ανάγκη να εγκαταλείπουν αυτοί οι άνθρωποι τις χώρες τους είτε για λόγους πολέμου είτε για οικονομικούς λόγους γιατί αναγκάζονται να φύγουν για να επιβιώσουν. Το 40% αυτών που ζητούν άσυλο στην Ευρώπη προέρχονται, μάλλον πηγαίνουν σε πέντε ε, χώρες της Ευρώπης. Τη Γαλλία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι τρεις από αυτές. Και πιστεύω ότι η αύξηση των αριθμών των προσφύγων για το 2014 είναι προφανής και οφείλεται κυρίως σε αυτά τα αποτρόπια γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στο Ιράκ και στη Συρία. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε υπεύθυνοι όλοι, ότι πρέπει να δείξουμε αλληλεγγύη και ότι οπωσδήποτε θα πρέπει να έχουμε μια κοινή πολιτική στο νότιο τμήμα της Ευρώπης και στο Βόρειο. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί η έκκληση της Λαμπεντούζα είχε πολύ θετική ανταπόκριση από μέρους των πολιτών μας. Δεν είναι μόνο παράνομοι αυτοί που έρχονται. Και σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε έναν μετανάστη σαν παράνομο. Βλέπετε τους αριθμούς ε, των θανάτων, η κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή. Πρέπει να μιλήσουμε περισσότερο για αυτήν την τρομερή καταστροφή που λαμβάνει η χώρα πολύ κοντά στην Ευρώπη. Είμαστε υπεύθυνοι και πρέπει να δείξουμε την αλληλεγγύη μας προς όλους αυτούς τους ανθρώπους που σήμερα υποφέρουν δίπλα στην Ευρώπη. Δεν μπορούμε να οικοδομήσουμε έναν ψηλό τείχο. Όσο θα υψώνουμε τείχη, τόσο θα αυξάνουμε τα προβλήματα. Πρέπει να υιοθετήσουμε λοιπόν ένα αλληλέγγυο μοντέλο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Συμφωνώ με όλα όσα ακούστηκαν. Την προηγούμενη εβδομάδα διοργάνωσα μια συνέντευξη τύπου με θέμα τη Λαμπεντούζα. Τα νούμερα που έχουμε είναι τρομερά ανησυχητικά. Από το 2008 υπήρξαν πάνω από 20.000 νεκροί στη Μεσόγειο. Μα γίνεται νεκροταφείο αυτή η θάλασσα πλέον. Την ίδια ώρα διαπιστώνουμε ότι η υπηρεσία Frontex δεν προσφέρει ικανοποιητικές λύσεις. Έλεγχος στα σύνορα, κάτι που δημιουργεί ένα φρούριο στην Ευρώπη. Δεν ανταποκρίνεται όμως στις ανάγκες των προσφύγων και των μεταναστών, είτε πρόκειται για άτομα που ζητούν πολιτικό άσυλο, είτε πρόκειται για οικονομικούς μετανάστες. Τι μπορεί να κάνει σήμερα ένας Ιρακινός, ένας Σύριος, ένας Λίβιος, ζει σε μια χώρα με την οικογένειά του που υπάρχει πόλεμος. Τι θα κάνατε εσείς και εγώ να προστατεύσουμε το Ελντοράντο της Ευρώπης. Ναι, τι μπορεί να κάνει η Frontex όμως με περισσότερες αρμοδιότητες και βλέπουμε την Ιταλία που είναι ο αποδιοπομπαίος τράγος. Εγώ πήγα στην Ελλάδα και ανησυχώ πάρα πολύ με τον ε, νέο επίτροπο από την Ελλάδα. Έχετε επισκεφτεί τα κέντρα κράτησης. Πρόκειται για εφιάλτη. Εγώ όταν ήμουν στην Ελλάδα ζήτησα να πάω στα κέντρα κράτησης. Μου είπαν όχι, απαγορεύεται. Γιατί οποιοδήποτε μπορεί να πάει να επισκεφτεί τις φυλακές στην Ελλάδα, παραδείγματο χάρη. Αν λοιπόν εμείς είμαστε υπέρ τη προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα πρέπει να έχουμε πρόσβαση στα κέντρα κράτηση. Εγώ διάβασα τις εκθέσεις της Amnesty International. Η κατάσταση είναι δραματική, φρικιαστική. Αυτός που πήγε και έμεινε τρία χρόνια στη Λαμπεντούζα διαπίστωσε ότι τα κοινοτικά κονδύλια χρησιμοποιούνται μέσω των εθνικών αρχών. Υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι που χρησιμοποιούν αυτά τα χρήματα. Ο κάθε μετανάστης έχει δικαίωμα για 35 ευρώ την ημέρα. Δίνονται αυτά τα χρήματα και τι έλεγχος γίνεται. Εμείς σαν Ευρωπαίοι βουλευτές δεν μπορούμε να δεχτούμε το έσχος αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα. Και στην Ιταλία ενδεχομένως. Δεν υπάρχει νοσοκομείο στη Λαμπεντούζα, παραδείγματο χάρη. Τώρα, όσον αφορά την αλληλεγγύη. Μόλις μάθαμε ότι θα δεχτεί 8.000 Ιρακινούς η Σουηδία. Μα αυτό είναι πραγματική αλληλεγγύη. Η κάθε χώρα πρέπει να πει πόσους πολιτικούς πρόσφυγες μπορεί να υποδεχτεί. Κανείς δεν κάνει τίποτα για να αυξηθούν οι αρμοδιότητες της Frontex χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη των κρατών μελών. Ας μας πει λοιπόν η Επιτροπή ποιος δεν θέλει να αυξήσει τις αρμοδιότητες της Frontex. Δεν μπορεί η Frontex απλώς να ελέγχει τα σύνορα. Πρέπει να σώνονται και ζωές. Και βεβαίως θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα κράτη-μέλη αυτά που εμποδίζουν αυτή την αύξηση αρμοδιοτήτων της Frontex. Ευχαριστώ πολύ. Να δίνω τον λόγο για τον κύριο Κυρκός. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι πραγματικά μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση και θα ήθελα να προσθέσω και εγώ την Ελλάδα σε όσα ε, ακούσαμε από τους προηγούμενους ομιλητές. Ήθελα όμως να τονίσω ότι δεν πρέπει να μείνουμε σε μια καταδίκη. Οι καταδίκες είναι σημαντικές αν συνοδεύονται και από τρόπους όπου το πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι εκατομμύρια άνθρωποι σειραίων προς την Ευρώπη δεν μπορεί η Ευρώπη να υποδεχθεί όλα τα εκατομμύρια των ανθρώπων τα οποία έχουν πρόβλημα από τις εμπόλεμες ή άλλες ζώνες κινδύνου. Είμαστε υπέρ μιας πολιτικής η οποία πρέπει να υλοποιήσει ε, το σύστημα του ασύλου στη βάση της αλληλεγγύης, μια πολιτική η οποία πρέπει να προσδιορίσει το θέμα της νόμιμης μετανάστευσης αναφερόμενη σε οικονομικούς μετανάστες και πρέπει να λάβει μέτρα ώστε αυτές οι πολιτικές να υλοποιηθούν. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο παίρνει και χρόνο. Αυτό που ζητάμε άμεσα είναι αυτή την αλληλεγγύη να την εκφράσουμε στην πράξη και στη Λαμπεντούζα και στα ελληνικά νησιά που μιλάμε για νησιά 100 ανθρώπων που έχουν 300 μετανάστες αυτή τη στιγμή, 300 ανθρώπους που έχουν βγάλει από τη θάλασσα, αυτή η αλληλεγγύη πρέπει να εκφραστεί πριν από το χειμώνα. Πρέπει να εκφραστεί αμέσως. Είναι ζητήματα τα οποία δεν μπορούν να τα παραπέμψουμε στις σωστές πολιτικές που θα υλοποιηθούν. Σε αυτή την κατεύθυνση θα θέλαμε να επαναφέρουμε την ερώτηση που κάναμε στον Επίτροπο, υποψήφιο Επίτροπο κύριο Αβραμόπουλο για να μην περνάνε οι άνθρωποι τη θάλασσα με τους δουλέμπορους, ε, αν θα μπορούσε να γίνει η αίτηση του ασύλου ή η αίτηση της α, μετανάστευσης σε τουρκικό έδαφος. Εμείς έχουμε την τύχη να έχουμε απέναντι στις αψακτές μας ένα οργανωμένο κράτος, έχουμε ήδη συμφωνίες μαζί τους. Αν θα μπορούσαν αυτές οι αιτήσει να γίνουν σε ε, μέρη που υπάρχει ε, επιτροπή από την Ευρωπαϊκή Ένωση που να τα εξετάζει αυτά ώστε να μην περνάνε τη θάλασσα, να μην μπαίνουν στο ρίσκο της παρανομίας. Και εδώ θα ήθελα να κάνω μια μικρή υποσημείωση. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι περνάνε τη θάλασσα πρόσφυγες. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι περνάνε τη θάλασσα άνθρωποι που διώκονται στις χώρες τους. Στην Ελλάδα υπάρχει ένα τεράστιο κύκλωμα το οποίο προωθεί ανθρώπους μέσα από τους σκλαβέμπορους, τους προωθεί κατευθείαν στην παράνομη εργασία, τους προωθεί κατευθείαν σε κέντρα τα οποία λυπάμαι που η λέξη έχει γίνει παγκόσμια αλλά θυμίζουν τη μαφία και αυτό είναι κάτι που κάνουμε πως δεν το καταλαβαίνουμε. Πρέπει να έχουμε σαφείς κανόνες, αλλά αυτοί οι σαφείς κανόνες πρέπει να είναι πραγματικοί και να εστιάζουν στην πραγματικότητα και όχι δυστυχώς μόνο σε έναν ανθρωπισμό ο οποίος δεν παίρνει καθόλου υπόψη ότι υπάρχουν τεράστια συμφέροντα που αυτή τη στιγμή κινούνται προς την Ευρώπη τελειώνω τώρα την κουβέντα είχαμε προχθές επειδή εμείς είμαστε δυστυχώς σε μια χώρα που δέχεται τους πρόσφυγες και τους μετανάστες δεν έχουμε τους 80.000 της Σουηδίας γιατί η ελληνική πολιτική είναι να κλείνουμε τα μάτια και να μην δίνουμε άσυλο όμως έχουμε πολύ περισσότερες χιλιάδες από ανθρώπους τους οποίους φιλοξενούμε τους οποίους εκμεταλλευόμαστε σε ένα μεγάλο βαθμό τους οποίους δεν θέλουμε να βλέπουμε οι οποίοι όμως ζουν στις γειτονιές μας αλλάζουν τη σύσταση των πόλεων δημιουργούν μια τεράστια σύγκρουση με τους κατοίκους. Είχα μια συνάντηση σε τέτοιες γειτονιές και η προσπάθεια είναι με, να μην κλείνουμε τα μάτια στο πρόβλημα, είναι εκρηκτικό και αν ακολουθήσουμε τη λογική που λέει δεν υπάρχουν ευρωπαϊκά σύνορα, το πρόβλημα δεν θα είναι απλά εκρηκτικό, το πρόβλημα θα σκάσει στα χέρια μας και η Ευρώπη δεν θα είναι πια η ίδια. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Now the floor... Τώρα, η κυρία Νταλή έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ξεκινήσω με κάτι που άκουσα εδώ η Μεσόγειος έχει γίνει νεκροταφείο. Ναι, γίνεται νεκροταφείο η ε, Μεσόγειος και εγώ που έρχομαι από τη Μάλτα είναι κάτι το οποίο μου είναι εξαιρετικά επώδυνο. Εγώ μεγάλωσα σε αυτό το νησί βλέποντας γύρω μου την ε, Μεσόγειο η οποία τώρα γίνεται κημητήριο ανθρώπων αλλά και κημητήριο ελπίδων. Θα πρέπει οπωσδήποτε ε, να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς να βρουν ένα νέο μέλλον και όχι να χάσουν τη ζωή τους ε, στη Μεσόγειο. Εγώ προέρχομαι από μια πολύ μικρή χώρα ε, που όμως αποτελεί σημείο εισόδου για αυτούς τους μετανάστες που βεβαίως είναι θύματα της παράνομης μετανάστευσης ε, γιατί ε, είναι γεγονός ότι το οργανωμένο έγκλημα και διάφοροι και κλπ εκμεταλλεύονται τους ανθρώπους αυτούς. Δεν τους δίνουν καν ούτε πλοία τα οποία να μην είναι πιο κάραβα και να μπορούν να τους ε, φτάσουν στην άλλη πλευρά της Μεσογείου οι άνθρωποι ε, οι οποίοι ζουν στη Μάλτα ή στη Λαμπεντούζα ή στα νησιά της Ελλάδας ή στην Ιταλία πιέζονται πάρα πολύ, τους ασκείται τεράστια πίεση και έχουν αφαιθεί στην τύχη τους, μόνοι τους εντελώς για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα αυτό. Ε, και σαν Ευρωπαϊκή Ένωση ε, σαν ε, ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και αυτούς τους ανθρώπους, τους πολίτες οι οποίοι αισθάνονται ότι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν μόνοι τους πλέον αυτό το, πρόβλημα και που είναι ένα θέμα που τους δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλη αγωνία. Ναι, βεβαίως το σημείο εισόδου είναι οι χώρες της Μεσογείου, αλλά το ζήτημα δεν είναι της μίας ή της άλλης χώρας, είναι ενωσιακό ζήτημα. Δεν είναι πρόβλημα ε, της μίας ή της άλλης χώρας ε, ή των νοτίων χωρών στο σύνολό τους. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο αφορά το σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να δράσουμε τώρα γιατί διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να αποφύγουμε και άλλες τραγωδίες στη Μεσόγειο. Τραγωδίες με πρωταγωνιστές ανθρώπους οι οποίοι φεύγουν από τις χώρες που προσπαθούν να βρουν ένα καλύτερο μέλλον ή την ασφάλεια. Ε, κινείται η task force ε, της ε, Μεσογείου από ό,τι ακούω και χαίρομαι που το ακούω αλλά κινείται πραγματικά με πάρα πολύ αργό ρυθμό. Θα πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες γιατί πραγματικά και εμείς αλλά και ο κόσμος που ζει στην Νότια Ευρώπη δεν την βλέπει την πρόοδο αυτή, δεν την βλέπει την κίνηση αυτή. Ε, μου λέτε πρέπει να αντιμετωπίσουμε το λαθρεμπόριο γενικά. Φυσικά στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ ε, συζητήσαμε και για την, ε, το, την υπηρεσία ΕΑΣΟ, συζητήσαμε και για το οργανωμένο έγκλημα. Πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπιστούν όλα τα ζητήματα αυτά. Θέλουμε λύσεις, όχι μόνο κάθε φορά που έχει προκύψει μια τραγωδία να λέμε δύο-τρεις κουβέντες και μετά να το ξεχνάμε. Ζητούμε μακροχρόνιες λύσεις ε, μιλάμε για την Frontex, αλλά η Frontex τελικά δεν αποτέλεσε λύση. Έχουμε τώρα την Frontex Plus. Ακούμε ότι 1η Νοεμβρίου ε, θα ε, ξεκινήσει και το Triton. Εντάξει, εγώ το δέχομαι, αλλά δεν έχουμε την απαραίτητη πληροφόρηση. Πρέπει να δούμε τι θα αποτελέσει ακριβώς το αυτό το Triton, πόσα χρήματα θα δοθούν. Θα πρέπει να ξέρουμε ακριβώς τι θα γίνει. Άκουσα και τον ε, ε, Επίτροπο που έλεγε ότι ο Τράιτον δεν θα είναι μονάχα ένας συνοριακός έλεγχος, θα είναι μια πολύ γενικότερη, συνολικότερη επιχείρηση. Εγώ κάνω μια έκκληση. Ε, λύσεις Τώρα πρέπει να καθίσουμε όλοι μαζί έτσι ώστε να βρούμε από κοινού λύσεις και έτσι ώστε και αυτοί οι άνθρωποι που ζουν σε αυτή την άκρη της Ευρώπης να μην αισθάνονται εντελώς εγκαταλελειμμένοι και να λένε ότι είναι δυστυχία που τελικά η ε, τύχη τους έφερε να ζουν στη Μεσόγειο. Κάτι πρέπει να γίνει άμεσα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Ε, Εύη Ελεονόρα, ο Μαριάς, ε, κυρία Μίση και η Σολεδάδ. Μπορώ να κλείσω τη λίστα των ομιλητών. Πρέπει ούτως ή άλλως να την κλείσουμε γιατί μετά έχουμε και άλλες αναφορές με παρουσία των αναφερομένων. Ελεονόρα. Ευχαριστώ. Να μην λησμονούμε ότι έχουμε και ένα άλλο παράγοντα που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας η συνθήκη του Δουβλίνου θα πρέπει να αναθεωρηθεί, θα πρέπει να ξεπεραστεί. Δεν είναι δυνατόν να βαραίνει πάντα την χώρα εισόδου ε, ε, ε, η διαχείριση, η διαχείριση ολόκληρου του ζητήματος και του προβλήματος. Είναι γεγονός ότι η κατάσταση πλέον έχει ξεφύγει, είναι τραγωδία και αφορά όλες τις χώρες της Νότιας Νότιας Ευρώπης. Ε, χώρες όμως οι οποίες ήδη ε, διανύουν ιδιαιτέρως χαλεπούς καιρούς από οικονομική άποψη. Δηλαδή ε, πέρα από την διαφορά την οικονομική μεταξύ Βορρά και Νότου έχουμε τώρα και αυτό το μεγάλο πρόβλημα το οποίο προστίθεται στη Νότια Ευρώπη. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να ξαναθυμηθούμε αυτά που οι πατέρες ιδρυτές ε, έλεγαν ότι πρέπει να γίνουμε μία ένωση. Θα πρέπει να μιλήσουμε όχι μόνο για ένωση πλέον αλλά και για κοινότητα, για κομινιτέ, ε, για μια κοινή επομένως διαχείριση των προβλημάτων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μαριάς παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, το θέμα που συζητούμε είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν αφορά μόνο την ε, Ιταλία, την Λαμπεντούζα, αφορά όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως αφορά τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου. Έχουμε χιλιάδες πρόσφυγες αλλά και χιλιάδες παράνομους οικονομικούς μετανάστες οι οποίοι επιδιώκουν να εισέλθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά το επιδιώκουν αυτό κυρίως από τις χώρες του Νότου, κυρίως από την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία. Επομένως αυξάνεται η πίεση των ροών αυτών στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου πρέπει να λάβετε υπόψη ταυτόχρονα ότι όλες οι χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου πλήττονται από ανεργία, από φτώχεια. Ιδίως δε η Ελλάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μια τεράστια ανθρωπιστική χρήση λόγω των καταστροφικών συνεπειών του μνημονίου που της έχει επιβληθεί σε αυτή την ανθρωπιστική κρίση προστίθεται και η νέα ανθρωπιστική κρίση που έχουμε με τα εκατομμύρια με τις χιλιάδες ε, πρόσφυγες και παράνομους μετανάστες που έρχονται στην Ελλάδα. Λέμε λοιπόν ότι η Ελλάδα δεν αντέχει άλλους παράνομους μετανάστες. Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλους ε, οι οποίοι έρχονται ως πρόσφυγες και ζητούν άσυλο. Είναι τεράστιος ο αριθμός και θα πρέπει να γίνει επίσκεψη και στην Ελλάδα όπως και στη Λαμπεντούζα για να δείτε την πραγματική εικόνα. Μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Επομένως πρέπει να έχουμε σοβαρά μέτρα αλληλεγγύης. Δηλαδή και τελειώνω με αυτό κυρία Πρόεδρε. Πρέπει να αλλάξει το Δουβλίνο 2 και πρέπει να πάμε σε μια ρύθμιση όπου οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανάλογα με τον πληθυσμό, την οικονομική τους κατάσταση και την έκταση να πάρουν τον αριθμό των παράνομων μεταναστών ή και των προσφύγων που ζητούν άσυλο. Δεν μπορεί να φορτώνονται δυστυχώς μόνο στην Ελλάδα, στην Ιταλία και σε άλλες χώρες. Εκεί πρέπει να κατευθυνθούμε για να δώσουμε μια λύση και αυτή τη λύση θα τη δώσουμε με μια ενιαία πολιτική στα ζητήματα αυτά. Thank σας ευχαριστώ, κυρία Μίτση. Ευχαριστώ. Πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο μας απασχολεί εδώ και χρόνια. Και δεν είδαμε βελτίωση ή και αποτελέσματα τέτοια τα οποία να αντικατοπτρίζουν τις συζητήσεις που έχουν γίνει για το θέμα αυτό. Θυμάμαι πριν από ένα χρόνο στο Στρασβούργο και σαν να ήταν χτες την Σεσίλια Μέστρομ που ε, ήρθε να μας μιλήσει μετά ε, ε, έχοντας επισκεφθεί την Λαμπεντούζα. Ήταν άσπρη, άσπρη πραγματικά σαν το χαρτί γιατί είχε δει φέρετρα παιδιών, φέρετρα με παιχνίδια πάνω τους. Έγινε κάτι. Όχι. Συζητούμε ξανά και ξανά τα ίδια πράγματα. Ας πούμε, δεν συζητάμε κάτι μακροπρόθεσμο και το οποίο θα αναζητήσει και τα πολλά δις τα οποία δίνει ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση σε χώρες της Αφρικής ας πούμε. Να αναζητηθούν τα χρήματα αυτά. Έχουν βοηθήσει για την δημιουργία υποδομών, έχουν βοηθήσει για την ε, στήριξη των ανθρώπων που ζουν στις χώρες αυτές έτσι ώστε λιγότερο να αισθάνονται την ανάγκη να εγκαταλείψουν τις χώρες αυτές εμείς ε, προσπαθούμε βεβαίως να δούμε με ποιο τρόπο ασφαλώς, με ασφάλεια δηλαδή μπορούν να περάσουν την ε, Μεσόγειο και πολύ σωστά το κάνουμε. Ε, ο, ωστόσο η Μάλτα ας πούμε είναι μια μικρή χώρα, είναι πάρα πολύ μικρή χώρα και μάλιστα νησιωτική. Ε, οι άνθρωποι αυτοί που ε, φτάνουν στη Μάλτα δεν θέλουν να μείνουν στη Μάλτα, θέλουν να πάνε στην Ευρώπη, στην, στην ε, υπηρετική Ευρώπη. Και βεβαίως δεν θέλουν δεν, δεν καταλαβαίνουν ότι κάποιοι πολίτες του νησιού αυτού ενδεχομένως ε, αισθάνονται ε, κάποια ρατσιστικά αισθήματα γιατί ε, αισθάνονται μία έλλειψη προσοχής, αισθάνονται μία έλλειψη ασφάλειας πλέον στις χώρες τους. Ναι, φυσικά έχω ακούσει και από πολλούς ανθρώπους την λέξη αλληλεγγύη αλλά παραμένει μία λέξη γιατί είναι κενή νοήματος πλέον η Ευρώπη θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα που αφορά και τις 28 χώρες. Και οι 28 χώρες θα πρέπει να καταλάβουν πόσο μεγάλο το πρόβλημα αυτό είναι. Και βεβαίως μετά από όλες αυτές τις καλές ε, λέξεις, αυτά τα καλά λόγια, τα ωραία και αφού έχουμε επιβιλήσει την καραμέλα της ελληνικής θα πρέπει κάτι να κάνουμε πλέον. Ευχαριστώ πολύ Σολεδάδα. Τελευταία ομιλήτρια. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι δεν είναι δυνατόν ε, να δεχτούμε λέξεις όπως απειλή για την ε, ύπαρξη των ε, υπολείπων, πρόβλημα κτλ. Ε, ξεχνούμε ότι μιλάμε για ανθρώπους. Ξεχνάμε ότι μιλάμε για κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Και βεβαίως εδώ δεν θέλουμε ούτε να ανοίξουμε τα σύνορα, ούτε να, να μην αντιμετωπίσουμε θέματα όπως είναι το τράφικινγκ ή όπως είναι το λαθρεμπόριο ή οτιδήποτε. Αλίμονο είναι θέματα τα οποία είναι εξαιρετικά πάρα πολύ σημαντικά, είναι εξαιρετικά σημαντικά, αλλά δεν πρέπει να συνεχίσουμε με αυτήν, σε αυτήν την ακινησία, σε αυτήν ε, την στάση που δεν μας οδηγεί πουθενά. Δεν μπορούμε να στρέψουμε το βλέμμα μας από την άλλη πλευρά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ασκήσει πλέον μια συνολική πολιτική, πολιτική η οποία θα βασίζεται στη συνεργασία όλων των χωρών, έτσι ώστε να μπορέσουν να βοηθηθούν και οι χώρες χώρες του Νότου για να αντιμετωπίσουν αυτά αυτό το πρόβλημα. Τα μέτρα είναι ανεπαρκή ε, και μην ε, ξεχνούμε ότι ε, όπως είπα και προηγουμένως πρόκειται για θέμα ανθρώπινο, πρόκειται εδώ για ανθρώπινα όντα και θα πρέπει όλοι μαζί να βοηθήσουν. Πριν από ένα χρόνο είχαμε την έκθεση για την ε, Λαμπεντούζα και είπαμε πολλά πράγματα, αλλά χρειάζεται ένα φόρουμ το οποίο θα αναλύσει το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι χώρες της Νότιας Ευρώπης. Μία ανάλυση σε βάθος η οποία θα μας επιτρέψει να αναλάβουμε πρωτοβουλίες σε πολιτικό επίπεδο. Η ΛΥΜΠΕ θα πρέπει να είναι η αρμόδια επιτροπή η οποία θα ε, ε, κάνει μια γνωμοδότηση, θα πρέπει δηλαδή να κάνει μια γνωμοδότηση έτσι ώστε να δούμε ποια μέτρα συγκεκριμένα μπορούμε να προτείνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ διαρκώς εργάζεται, είμαι συντονίστρια και πραγματικά επεξεργάζεται αυτά τα θέματα διαρκώς. Όσον αφορά την αλληλεγγύη, βεβαίως δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υποστηρίζουμε αυτήν την έννοια. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο συγκεκριμένα νομοθετικά κείμενα να βασιστούν στην αλληλεγγύη. Πρέπει σαφώς και να στηρίξουμε κάθε πρωτοβουλία για περισσότερη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Κάποιος συνάδελφος, δεν είναι όμως σήμερα εδώ, είπε ότι δεν μπορεί μόνο η Ελλάδα και η Ιταλία να αναλάβουν το βάρος όλων αυτών που ζητούν ε, άσυλο. Απ' την άλλη βλέπουμε ότι στην ε, Σουηδία πάνω από 80.000 άτομα ζήτησαν άσυλο φέτος. Τελικά η Σουηδία είναι αυτή που παίρνει το μεγαλύτερο αριθμό των πολιτικό άσυλο. Πρέπει λοιπόν να δούμε ότι σε αυτές τις καταστροφικές ε, ε, περιπτώσεις όπως 300 ε, άτομα που έχασαν τη ζωή τους στη Λαμπεντούζα, κάτι πρέπει να κάνουμε. Μόνο για το 2014 πάνω από 3.000 άτομα έχασαν ήδη τη ζωή τους στη Μεσόγειο. Πραγματικά λοιπόν η τραγωδία αυτή συνεχίζεται στη Μεσόγειο. Η μόνη λύση για να καταπολεμήσουμε όλους αυτούς τους δουλέμπορους και την παράνομη μετανάστευση είναι να θεσπίσουμε κάποιες ασφαλείς οδούς. Και πραγματικά ευχαριστώ πολύ την Επιτροπή για τη δήλωσή της και θεωρώ ότι και ο πρόεδρος της Επιτροπής της δηλώσεις του έχει αναγνωρίσει το πρόβλημα λέγοντας ότι είναι άμεσο και ότι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Η Επιτροπή Αναφορών τώρα πρέπει να συνεργαστεί με την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή, την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Έχετε εξάλλου και ένα πρωτόκολλο για την συνεργασία για θέματα μετανάστευσης και όπως ξέρετε η έκθεση για το θέμα αυτό της Amnesty International δημοσιεύεται σήμερα. Εμείς λοιπόν σαν πολιτικοί αλλά κυρίως σαν άνθρωποι, σαν Ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όλα αυτά και να πούμε ότι πραγματικά η Ευρώπη ήταν χώρος από τον οποίο έφευγαν άνθρωποι και μετανάστευαν πριν από έναν αιώνα. Και 25% του πληθυσμού μας είχε μεταναστεύσει. Σήμερα η Ευρώπη είναι ένας ε, τόπος στον οποίο έρχονται οι πρόσφυγες και οι μετανάστες. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι εν δυνάμει μετανάστης είναι ο καθένας από μας. Υπάρχουν περιοχές στις οποίες σήμερα υπάρχει πόλεμος και οι άνθρωποι που μένουν εκεί εγκαταλείπουν τα σπίτια τους, τις χώρες τους. Εμείς λοιπόν σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σαν Επιτροπή Αναφορών πρέπει να συνεργαστούμε με την Επιτροπή, με το Συμβούλιο, με τις αρμόδιες επί της επιτροπές, με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ δηλαδή, για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα φαινόμενα. Θα σας δώσω το λόγο, Ματίας, για να ολοκληρώσετε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας υποστηρίξω για όλα όσα είπατε. Ήταν πάρα πολύ ουσιαστική η συζήτηση. Έχουμε μπροστά μας πολιτικές προκλήσεις και σαφώς χρειάζεται οριζόντια προσέγγιση και αντιμετώπιση. Για όλους όσους θέλουν περισσότερες πληροφορίες, με μεγάλη χαρά μπορώ να στείλω στη Γραμματεία της Επιτροπής Αναφορών ε, την δάση μας για τη Μεσόγειο και θα ήθελα επίσης να πω ότι το Δεκέμβριο ολοκληρώσαμε τις εργασίες μας στην Task Force για την ε, Μεσόγειο. Συνεργαζόμαστε όμως σήμερα με την Ιταλική Προεδρία. Την Παρασκευή η Ιταλική Προεδρία θα παρουσιάσει την έκθεσή για το θέμα αυτό. Όσον αφορά τώρα τη χρηματοδότηση, μετά την Λαμπεντούζα πήραμε 10 εκατομμύρια ευρώ σαν Ιταλία για τις κατεπίουσες δράσεις. 7,9 ευρώ πήραμε για την ενίσχυση της Frontex και 12 εκατομμύρια ευρώ για τον επαναπατρισμό. Συν 13 εκατομμύρια ευρώ που είχαμε πάρει πέρσι. Ο κύριος Μποργκέζο είπε ότι υπάρχει και ο φόβος της εγκληματικότητας η οποία αυξάνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήθελα να σας πω ότι η καταπολέμηση όλων αυτών των παράνομων εμπορίων ανθρώπων είναι κάτι που θα ασχοληθεί και με αυτό το θέμα στο τέλος του μήνα στην Κατούμα υπό την αιγίδα της Ιταλικής Προεδρίας διοργανώνεται αυτή η συνάντηση και έχει σαν σκοπό να μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν αυτές οι δράσεις ε, από τα προγράμματα περιφερειακής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σαφώς και πρέπει να έχουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και αυτό σημαίνει, και αυτό δεν πρέπει να παραμείνει λόγια, η Frontex κάνει πολύ αποτελεσματική δουλειά. Έλεγχο των συνόρων και διάσωση ανθρώπινων ζώων. Και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συνεχίσουμε τη δράση μας σε όλους τους τομείς. Η Ελλάδα. Σήμερα δεν συζητούμε για την Ελλάδα, αλλά θέλω να σας πω ότι βεβαίως και είναι δυνατόν κάποιος να επισκεφτεί τα κέντρα κράτησης στην Ελλάδα. Η Επιτροπή πάει συχνά, έχουν πάει και κοινοβουλευτικές ε, αποστολές και έχουν επισκεφτεί τα κέντρα κράτηση στην Ελλάδα και είμαστε σε πολύ στενή επαφή με τη Μάλτα, τη Βουλγαρία και την Ελλάδα που είναι χώρες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Εκατομμύρια ευρώ έχουν δοθεί στις χώρες αυτές για να συνεχίσουν την αντιμετώπιση αυτών των ε, προσφύγων. Αναφερθήκατε και στην Τουρκία κάποιος από εσά. Αυτό όμως είναι θέμα που πρέπει να το αναλάβει η Γενική Διεύθυνση για την διεύρυνση. Η Τουρκία παρόλα αυτά κάνει πάρα πολλές προσπάθειες όσον αφορά την ενσωμάτιση και την προστασία πολλών προσφύγων που έρχονται από την Συρία. Να επαναλάβω επίσης ότι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά την ειδική κατάσταση της Μάλτας. 11 εκατομμύρια έχουν ε, δοθεί στη Μάλτα σαν έκτακτη βοήθεια. Κυρία Πρόεδρε, το 70% των αιτήσεων για άσυλο γίνονται στην Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Γαλλία και το Βέλγιο. Και τη Σουηδία, συγγνώμη σε αυτές τις πέντε χώρες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λέλη που εκπροσωπείτε εδώ όλους τους αναφέροντες. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω την Προεδρία της Ιταλίας, την Επιτροπή. Θεωρώ ότι πρέπει να κλείσουν αυτές οι αναφορές. Υπάρχουν πάρα πολλές άλλες που ασχολούνται ακριβώς με το ίδιο θέμα. Να πούμε λοιπόν ότι δεν ακούω τίποτα, αλλά προτείνω να τις κλείσουμε τις αναφορές. Λέτε ναι, το ΕΛΚ λέει ναι τουλάχιστον. Και μπορείτε αν θέλετε να εγκαταλείψετε την αίθουσα όσοι είστε εδώ για το σημείο 8 γιατί περνάμε τώρα στο σημείο 9. Η σοσιαλιστική ομάδα θα προτιμούσα να μείνει ανοιχτή για να δούμε ακριβώς πώς θα συνεργαστούμε με την ΛΥΜΠΕ και να δούμε ακριβώς και την έκθεση της Ιταλικής Προεδρίας. Ωραία. Θα κρατήσουμε αυτό το θέμα ανοιχτό. Και ίσως για σήμερα να έχουμε και πολλές αναφορές που αφορούν τα ίδια θέματα από άλλους αναφέροντες. Οπότε προτείνω να κλείσουμε αυτές οι συγκεκριμένες αναφορές. Δηλαδή του κυρίου Λέλη ας πούμε ο οποίος ήρθε και του δόθηκαν απαντήσεις στο μέτρο του δυνατού. Μπορούμε και για αντίστοιχες αναφορές να κάνουμε το ίδιο. Μάλλον ναι, λέτε έτσι. Όχι. Κοιτάξτε, σε καμία περίπτωση δεν κλείνει το θέμα Λαμπεντούζα ή αυτών που ετούν άσυλο. Απλώς κλείνουμε αυτήν τη συγκεκριμένη, αυτές τις αναφορές τις οποίες συζητήσαμε σήμερα. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές άλλες με ίδιο αντικείμενο οι οποίες είναι πιο ενημερωμένες, αν θέλετε, πιο επίκαιρες. Αυτές είναι παλιές, ας τις ξεφορτωθούμε με την έννοια ότι θα μπορέσουμε να ασχοληθούμε με άλλες αναφορές για την Ισπανία, για τη Λαμπεντούζα και δεν ξέρω πού αλλού. Αλλιώς θα πρέπει να παραμείνουμε με αυτές τις αναφορές ανοιχτές. Συμφωνείτε τελικά. Είπατε προτείνεται ορθά να ε, κλείσουμε την αναφορά ε, αυτήν την ε, αναφορά του κυρίου Λέλη, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν άλλες σχετικές με πολλά ζητήματα που εκκρεμούν ακόμα. Γιατί, κοιτάξτε, εάν κλείσουμε τότε θα εξακολουθήσουμε να έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Δηλαδή συζητούμε, συζητούμε, αλλά τελικά δεν καταλήγουμε σε καμία λύση και σε καμία τελική πρόταση. Ναι, ε, μπορώ να συμφωνήσω μπορώ να συμφωνήσω. Γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να κάνουμε και μια συγκεκριμένη πρόταση, κάποια συγκεκριμένη πρωτοβουλία, τι θα κάνουμε. Είπαμε, προτείναμε συνεργασία με την ε, ΛΥΜΠΕ, δεν έγινε τίποτα. Συνεργασία με την Ελληνική Προεδρία. Κοιτάξτε, ε, ε, να δούμε πρώτα αν μπορούμε να κάνουμε κάτι συγκεκριμένο και μετά να αποφασίσουμε αν θα κλείσουμε ή αν δεν θα κλείσουμε. Mrs. Συμφωνώ απολύτως με αυτά που μόλις είπε η συνάδελφος. Κοιτάξτε, ε, είπαμε ότι αυτές οι αναφορές θα πρέπει να είναι ε, μαζί. Η διαδικασία, τη διαδικασία την είχαμε συζητήσει. Αν πρόκειται να αλλάξουμε διαδικασία θα πρέπει να το, συζητήσουμε στους ε, συντονιστές. Νομίζω ότι θα πρέπει να δοθεί συνέχεια, αν μη τι άλλο. Τώρα, εάν έχει αλλάξει κάτι στη διαδικασία να μας το πείτε, αλλά δεν νομίζω ότι έχει γίνει κάτι τέτοιο εδώ. what, what I'm trying to say... Αυτό που προσπαθώ να πω, λέει η Πρόεδρος, είναι ότι έχουμε τόσες πολλές αναφορές με το ίδιο ακριβώς θέμα που, θα, που έρχονται ε, αργότερα, που δεν έχει έννοια να αφήσουμε αυτή τη συγκεκριμένη ανοιχτή καμία έννοια. Εάν βεβαίως επιμένετε μπορούμε να την ανοίξουμε. Θέλετε να ξαναβάλουμε το, τις ε, αναφορές αυτές ξανά για μία ακόμα φορά ε, στην ε, ημερήσια διάταξη. Ούτως ή άλλως ένας από όλους αποφάσισε να είναι παρόν. Οι υπόλοιποι δεν ήρθαν καν. Πίτερ. Καταλαβαίνω τι λέει η, συγε η πρόεδρος, συγγνώμη. Υπάρχει και ένας συμβιβασμός. Δηλαδή, να τις αφήσουμε ανοιχτές, αλλά να μην είμαστε υποχρεωμένοι οπωσδήποτε να τις ξαναεπεξεργαστούμε. Αν προκύψει κάτι, μπορούμε να το κάνουμε. Τις αφήνουμε ανοιχτές, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι να επανέλθουμε και να τις ξαναεπεξεργαστούμε. Θα αποφασίσουν οι συντονιστές για το τι μελιγενέστε με αυτές τις αναφορές. Γιατί μπορούμε κάλλιστα είτε να τις κλείσουμε είτε να τις αφήσουμε ανοιχτές, αλλά να πούμε ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει υποχρέωση να επανέλθουμε σε αυτές. Δεν ξέρω, σας ε, αρέσει αυτή η συμβαστική πρόταση. Έχω την εντύπωση ότι δεν υπάρχει μεγάλη διαφωνία. Όλοι θέλουμε να προχωρήσουμε στην επεξεργασία επόμενων αναφορών, έτσι δεν είναι. Νομίζω ότι όλοι πήρατε τις πληροφορίες από την Επιτροπή. Συζητήσαμε, ήρθαν εδώ οι αναφέροντες. Τώρα, αν θέλετε να την αφήσουμε ανοιχτή, ποτέ δεν θα μπορέσουμε να επεξεργαστούμε τις εκατοντάδες των αναφορών που περιμένουν και τις οποίες δεν έχουμε χρόνο να επεξεργαστούμε. Τι να σας πω. Αν επιθυμείτε παρόλα αυτά να παραμείνουν ανοιχτές, θα τις αφήσουμε ανοιχτές. Εκτός από αυτή του κυρίου Λέλη. Και θα δούμε αν υπάρχει άλλος τρόπος επεξεργασίας, με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, με την Προεδρία αυτή και τις επόμενες, γιατί θεωρώ ότι αυτά τα θέματα θα τα βρούμε μπροστά μας στο μέλλον. Αν θέλετε να παραμείνουν ανοιχτές αυτές οι ε, αναφορές, θα το κάνουμε. Εγώ προσωπικά θα ήμουν υπέρ του να τις κλείσουμε, γιατί επαναλαμβάνω υπάρχει πληθώρα αναφορών για παρόμοια και ίδια θέματα πάρτε μία απόφαση γιατί κάπως πρέπει να συνεχιστεί η εργασία αυτής της Επιτροπής. Ανοιχτές, ωραία, εκτός από αυτή του κυρίου Λέλη. Και τώρα περνάμε σε θέματα περιβάλλοντος, στο σημείο 9, με πολλά, πολλά θέματα, πολλές αναφορές. Θα δούμε μάλιστα και το βίντεο Βιντάλ Μαρτίν. Είστε εδώ? Ναι.

είχαμε το θαλάσσιο οικοσύστημα στην περιοχή των Κανάριων νήσων το οποίο απειλείται από, τις, από το ενδεχόμενο εξορίξεων. Αλλά δυστυχώ ο ήχο από το βίντεο είναι πολύ κακή ποιότητα και δεν μπορούμε να το μεταφράσουμε. La SECAC ha participado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 ναι, ε, πρέπει να πούμε ότι ήταν ε, δυστυχώς ε, άσχημος ο ήχος, δεν μπόρεσαν οι διερμηνείς να το μεταφράσουν. Παρακαλώ, η Κάρμεν έχει το λόγο. Πού είστε, Κάρμεν? Καλώς ορίσατε. Καλώς ορίσατε, σας δίνω το λόγο αμέσως. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους κυρίους και τις κυρίες βουλευτές που μας ακούν για άλλη μια φορά για ένα θέμα που είναι τόσο σημαντικό όχι μόνο για τα Κανάρια νησιά και όχι μόνο για το Ισπανικό κράτος αλλά για ένα θέμα παγκόσμια σημασίας. Θέμα που αφορά και τη δημοκρατία γιατί λέμε ότι η, η κοινωνία των Καναρίων επανελειμμένος από το Μάρτι του 12 και μετά βγήκε μαζικά στο, στους δρόμους και το 2014 πάλι είχαμε πολλές διαδηλώσεις για να εκφράσουμε την διαφωνία μας με αυτό το σχέδιο εξορίξεων και τον Ιούνιο σε 7 του Ιούνιου φέτος, μια εβδομάδα μετά από την υιοθέτηση της δήλωσης μάλλον της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την Ισπανική κυβέρνηση, πάλι βγήκαν στα Κανάρια στους δρόμους πάνω από 300.000 άτομα. Οι δημόσιες αρχές των Καναρίων, το τοπικό κοινοβούλιο παντλημένος, υιοθέτησε αυτή την απόρριψη, ζητώντας από την κυβέρνηση να σταματήσει αυτή τη διαδικασία εξορίξεων για το πετρέλαιο στην Λαθαρότα και στην Φορτεβεντούρα. Και η τοπική κυβέρνηση των Καναρίων από τα 7 ίσια που εκπροσωπούνται στο τοπικό κοινοβούλιο και αυτό εξέφρασε την αντίθεσή του, όπως και η Δήμοι το ίδιο και κυρίως οι Δήμοι της Φορτεμετούλα και Λανθαρότε. Επίσης η διεθνής κοινότητα εξέφρασε την αλληλεγγύη της και έχουν τρομοκρατηθεί από τα σχέδια της Ισπανικής κυβέρνησης σε σχέση με την εξόρυξη πετρελαίου. Να σας πω ότι αυτό το θέμα ένα θέμα που ξεπερνά τα Κανάρια και το Ισπανικό κράτος ένα θέμα το οποίο αφορά όλους μας, γιατί μιλάμε για τον θαλάσσιο χώρο μέγιστης παγκόσμιας σημασίας όσον αφορά την παρουσία κοιτοδών και βιοπικιλότητας. Αυτό είναι άλλο ένα ζήτημα που θα θέλαμε να θίξουμε και θα θέλαμε να γνωρίζετε κάποια θέματα προκατακτικά. Τα Κανάρια νησιά βρίσκονται 4.000 χιλιόμετρα περίπου από τις Βρυξέλλες αποτελούν ένα τουριστικό προορισμό ισχυρό. Πάνω από δύο εκατομμύρια τουρίστες ετησίως. Επισκέπτονται πολλοί τουρίστες στα μέρη μας για να απολαύσουν από το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Δύο εκατομμύρια κάτοικοι είναι εκατομμύρια τουρίστες. Είναι όμως και ένα φυσικό μέρος της φυσικής παγκόσμιας κληρονομιάς. Έχουμε τέσσερα εθνικά πάρκα όπου θα πρέπει να προσθέσουμε 144 φυσικούς χώρους προστατευόμενους από τους ντόπιου νόμους. Πάνω από 44% της συνολικής επιφάνειας του αρχιπελάγου των Καναρίων ε, διέπεται από μέτρα προστασίας. Εξάλλου και το ίδιο το δίκτυο Natura περιλαμβάνει πολλές περιοχές ε, προστασίας στα Κανάρια. Επίσης υπάρχουν πάρα πολλά μέρη που έχουν κηρυχθεί παγκόσμια πολιστική κληρονομιά, Λαγκομέρα και άλλα νησιά, όπως και η Φορτεβεντούρα. Μιλάμε λοιπόν για ένα θέμα που έχει μέγιστη σημασία από την σκοπιά του περιβάλλοντος και από την σκοπιά της δημοκρατίας. Εάν δεν τηρηθεί, αν δεν γίνει σεβαστή η βούληση των πολιτών και η βούληση των επισήμων συγκροτημένων αρχών των τοπικών για την προστασία αυτής της φυσικής κληρονομιάς, η οποία ξεπερνάει κατά πολύ τους πολίτες που ζούμε εκεί, τους κατοίκους, οι οποίοι είμαστε απόλυτα ευτυχισμένοι που είμαστε σε θέση να έρθουμε εδώ, αλλά και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από τη διεθνή αλληλεγγύη γιατί τα τελευταία δύο χρόνια είπαμε βγήκαν στους δρόμους αλλά βγήκαν στους δρόμους και στις Βαλεαρίδες υπέρ των Καναρίων στη Βαλένθια, στην ε, Μαδρίτη, στη Βαρκελόνη, στον Μπιλμπάο, στη Σεβίλη, στο Λονδίνο, στο Παρίσι, στο Βερολίνο, στη Νέα Υόρκη Είμαστε λοιπόν ιδιαίτερα ευτυχισμένοι γι' αυτό. Αυτό το σχέδιο εξέρωξης που η κυβέρνηση της Ισπανίας, η κυβέρνηση του Λαϊκού Κόμματο ήθελε να σιωπήσει και η πολυεθνική Ρεψόλ, η οποία θέλει να καταστρέψει τις φυσικούς πόρους του νησιού, γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να το κρύψουν, να το αποκρύψουν και δεν μπορούν να λειτουργήσουν με τον ίδιο τρόπο που λειτουργούσαν δεκαετία του 90 όπου αυτή η πολυεθνική, και αυτό είναι τεκμηριωμένο, έκανε σοβαρέ, σοβαρότατε, μεγάλε ζημιέ στον Αμαζόνιο, στην Αργεντινή, στη Βολιβία, στον Σημερινό. Ξέρουν όμω ότι τα Κανάρια βρήκαν μια κοινωνία η οποία είναι πολύ δραστήρια και ξέρουν τα μέσα τι γίνεται και μας επέτρεψαν να εκφραστούμε και η Επιτροπή Αναφορών του Κοινοβουλίου μας επέτρεψε το ίδιο και οι διάφορες δραστηριότητες των τοπικών αρχών της και τοπικής κυβέρνησης όλοι μας κινητοποιηθήκαμε για να υποβάλουμε διάφορες αναφορές. Και επιτρέψτε μου τώρα να σχολιάσω κάποια σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις από το Γενάρη, από τις 21 του Γενάρη μέχρι σήμερα. Κάτι το οποίο αφορά την, την Κομισιόν. Κομισιόν που προσπάθησε να αποσιωπήσει αυτά που συνέβησαν από το Γενάρη μέχρι σήμερα. Τότε δεν είχαμε τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων το Γενάρη. Εμείς καταγγέλαμε το γεγονό ότι σε αυτή τη μελέτη περιβαλλοντικών ε, επιπτώσεων υπάρχει μη τήρηση του και μη εφαρμογή του, κοινοτικού, του βασικού κοινοτικού και εκτιμένου. Υπάρχει λοιπόν η μη τήρηση για τους εξή λόγους Και κύριοι και κυρίες ευρωβουλευτές πρέπει να γνωρίζετε ότι η Κομισιόν απέφυγε να ασχοληθεί ή να λάβει υπόψη ένα πολύ σημαντικό γεγονό. Το Μάρτι του 2013 η εταιρεία Repsol υπέβαλαν περιβαλλοντικές πληροφορίες σε ένα αρχικό έγγραφο, βάσει του οποίου η, η αρχή βιωσιμότητας των ακτών και η, η αρχή περιβαλλοντική επεξεργάστηκαν και συνέταξαν ένα έγγραφο περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Σε λιγότερες από 40 μέρες δόθηκε στη Ρεψόλα αυτό το έγγραφο. Σε λιγότερο από 40 μέρες ένα πολύ περίπλοκο έγγραφο περιβαλλοντικών επιπτώσεων δόθηκε στην ε, Ρεψόλ και υποβλήθηκε στη συνέχεια για δημόσια διαβούλευση στις 29 του Ιούλη ε, του 2013, σε λιγότερο από 40 μέρες. Απίστευτο αυτό. Πώς γίνεται, πώς γίνεται αυτό σε τόσες λίγες μέρες, σε τόσες λίγες μέρες να εκπονείται μια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και να δουλεύει κανείς για μια εταιρεία και όχι για το κοινό καλό. Είχαμε λοιπόν την μελέτη αυτή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και επιτρέψτε μου Πρόεδρε. Να συνεχίσω, επειδή υπάρχουν και πέντε αναφερόμενοι και το συζήτησαμε τη γραμματεία ώστε να συνοψίσουμε, να υπάρχει μια κοινή παρουσίαση που αφορά όλες αυτές τις αναφορές. Όπως σας παρακαλώ επιτρέψτε μου να συνεχίσω. Συμφωνείτε, μπορώ, μπορώ να συνεχίσω. Ευχαριστώ. Υποβλήθηκαν λοιπόν για δημόσια διαβούλευση. Πρέπει όμως να γνωρίζετε ότι η περίοδος της δημόσιας διαβούλευσης ήταν σύντομη. Το Φλεβάρι του 2014 η Γενική Διεύθυνση Οικολογικής Αξιολόγησης ζήτησε από τη Ρεψόλ νέα μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και επιπλέον 26 έγγραφα. Αυτό δεν το γνωρίζει η Κομισιόν. Αυτό η Κομισιόν το αγνοεί. Γι' αυτό λέει ότι έχει γίνει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία είναι καλή. Δεν το γνωρίζει αυτό η Κομισιόν. Το Φλεβάρι λοιπόν του 2014 η Γενική Διεύθυνση Αποτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ζήτησε από την ε, Ρεψόλ ένα κατάλογο 37 εγγράφων. Δεν το γνωρίζει επειδή την ε, ενημέρωσε η Ισπανική κυβέρνηση. Επίσης το Μάη μέσω από αυτή, τη, μέσα από αυτή την διεύθυνση μας ενημέρωσαν για έγγραφα που υποβλήθηκαν. Επίσης δεν γνωρίζει ότι η Γενική Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής μας ενημέρωσε για την ύπαρξη και άλλων εγγράφων. Τη στιγμή που η μελέτη χωρίς ε, διαβούλευση στην ουσία υιοθετήθηκε και αποτελεί αποτέλεσμα ενός προεδικού ενός διατάγματος που βγήκε με την πίεση της βιομηχανίας του πετρελαίου ιδιαίτερα για τα Κανάρια. Και πρέπει να ξέρετε, Πρόεδρε, ότι στην Φορτεβετόρα υπάρχει μεγαλύτερη παρουσία κοι, κοιτοειδών παγκοσμίω. 35%. Πρέπει να ξέρετε λοιπόν από το 2009 και μετά η Κομισιόν ζήτησε από την Ισπανική Κυβέρνηση να υποβάλει προτάσεις που να αφορούν το θαλάσσιο χώρο. Και πράγματι το 2009 ξεκίνησε η Ισπανική Κυβέρνηση να μελετά μέχρι το 2013 ένα νέο πρόγραμμα και υποβλήθηκαν εκεί διάφορα σχέδια και προτάσεις για χώρους συγκεκριμένου των Καναρίων. Το 2011 διάφορες επιστημονικές αρχές υπέβαλαν υπόμνημα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος λέγοντας ότι η αξία της βιοπικιλότητας αυτό το θαλάσσιο χώρο είναι τόσο μεγάλη που θα έπρεπε να διευρύνουν τη ζώνη προστασίας και αυτό είχε γίνει δεκτό το 11 από την Κομισιόν. Ξέρετε λοιπόν στις 16 ε, Μαρτίου του 2012 εγκρίθηκε το βασιλικό διάταγμα. Ο, ο κύριος Κανιέτο, ο υπουργός περιβάλλοντος τότε, έκανε τα στραβά μάτια και έχει, έχει ποινική ευθύνη. Πρέπει να το διερευνήσει αυτό η Κομισιόν γιατί υιοθετήθηκε αυτό το βασιλικό διάταγμα, δίνοντα άδεια για εξορίξει, χωρί χωρίς να ληφθούν υπόψη αυτά τα επιστημονικά στοιχεία. Γνωρίζοντα ότι τεράστιο ποσοστό που αφορά αυτέ τι εξορίξει βρίσκεται στον χώρο που λέγαμε προηγουμένω, στον προστατευόμενο. Όλα αυτά λοιπόν τα στοιχεία είναι πολύ ανησυχητικά. Αυτό σημαίνει, Πρόεδρε, ότι δεν μπορούμε να αποδεχτούμε εδώ την πρόταση μεριβαλλοντικών επιπτώσεων και την διαδικασία, διαδικασία εκτροπής του κοινωνικού καθολικού συμφέροντος. Σήμερα λοιπόν ζητάμε κάτι πολύ συγκεκριμένο πρόεδρε από εσάς που το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να παραβλέψει και ξέρω ότι υπάρχουν ευαισθησίες. Ζητάμε λοιπόν κάτι πολύ συγκεκριμένο. Λέμε εμείς, αν ο κύριος Κανιέτη ο οποίος ήταν υπουργός περιβάλλοντος στην Ισπανία. Αν ο κ. Κανιέτε λοιπόν ε, αντιμετωπίζει ένα ασυμβίβαστο για θέση του Επιτροπού λόγω συμφερόντων στον ε, τομέα του πετρελαίου μπορεί να αναγνωρίζει αυτή τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων όπως λαμβάνει υπόψη αυτά τα στοιχεία και την αντίδραση του ντόπιου πληθυσμού. Μπορεί να αποδέχεται όλη αυτή η διαδικασία που οδήγησε στην εξουσιοδότηση. Ξέρετε, Πρόεδρε, ότι σήμερα εκπνέει η προθεσμία σήμερα και ζητάμε, Πρόεδρε, η Επιτροπή Αναφορών του Κοινοβουλίου να απαιτήσει από την Κομισιόν να υιοθετήσει τα απαραίτητα μέτρα. Ε, εδώ δεν είμαστε να συζητήσουμε τον υποψήφιο επίτροπο, είμαστε εδώ για να συζητήσουμε αναφορά σα, κύριε Φερνάντεθ, λέει η Πρόεδρο. Ωραία, ωραία, ζητώ συγγνώμη αλλά αυτό έχει άμεση σχέση όλα αυτά που έγιναν τα δύο τελευταία χρόνια με αυτή τη δικασία για τον κύριο Κανιέτη. Αυτό είναι αναπόφευκτο, είναι η πραγματικότητα. Σας ζητώ να ολοκληρώσετε παρακαλώ, γιατί υπάρχουν και άλλοι ομιλητές στο κατάλογο μου. Συγχωρήστε με και ολοκληρώνω. Ζητάμε λοιπόν από την Επιτροπή Αναφορών να απαιτήσει από την Κομισιόν να εθετήσει μέτρα για την αναστολή αυτής της διαδικασίας, τη διερεύνηση των επιστημονικών στοιχείων και την άσκηση κοινοτικού, κοινοτικού ελέγχου ώστε να προστατευτούν αυτές οι περιοχές και εντωμεταξύ εν αναμονή των επιστημονικών στοιχείων που αφορούν τις εξορίξεις. Αν και πρέπει να δει επίσης η Κομισιόν κατά πόσο μπορούν να εφαρμοστούν αυτά που θέλει το Υπουργείο Μηχανής της Ισπανίας και αυτά που θέλει η Πολυεθνική Εταιρεία Repsol. Σα ευχαριστώ πολύ. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Έχω δύο βίντεο. Υπάρχει ένα της Νατάσα Αγγιγιάρ με διερμηνία, αν δεν κάνω λάθος. Ε, να προχωρήσουμε λοιπόν στο βίντεο αυτό αμέσως. Παρακαλώ. Hello, my name is... Γεια σας, λέγομαι Νατάσα Αγγιλάρ και εργάζομαι στο Διεθνός Κάμπους Αριστείας στα Κανάρια νησιά όπου διευθύνω ε, ακουστική έρευνα για τα κοιτόδια από το 2006 και εργάζομαι ε, σε μια υπηρεσία που μελετά το θαλάσσιο περιβάλλον στο αρχιπέλαγος ε, πάνω από 30 χρόνια. Πολύ πλούσιο περιβάλλον, πάνω από 7.000 θαλάσσια είδη, αυτό απορρέει και από την ανακήρυξη αυτή τη περιοχής ως ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχής από τον Διεθνή Αυθυλιακό Οργανισμό. Επίσης και ο πληθυσμός της ε, περιοχής παρουσιάζει ιδιαίτερα, εξαρτάται μάλλον από τα καθαρά νερά για την επιβίωση αυτών των ειδών. Έχουμε στην φορτευτό και λαθαρότητα μια προστατευόμενη περιοχή, 11 χιλιόμετρα μακριά δηλαδή, μόνο από το σημείο εξόριξη των σχεδίων τη Ρεψόλ. Και εδώ στο μπλε μπορεί να, βλέ, να δείτε αυτά τα μέρη που βρίσκονται τα κοιτόδη και άλλα θαλάσσια θαλαστικά. Αυτή όμως η δική περιοχή προστασίας ήταν πιο μεγάλη το 2011 και περιλάμβανε αυτή την διάμεση ζώνη η οποία ακριβώς επικαλύπτεται με τα σημεία εξόρυξης τώρα μειώθηκε αυτή η, περιοχή η προστασίας και δεν ξέρουμε αν έγινε ακριβώ λόγω αυτών των σχεδίων εξόρυξης. Η περιοχή αυτή είναι πάρα πολύ ε, πλούσια ε, σε ε, βαθιά και ρηχανερά. νερά. Υπάρχουν κοράλια και κοραλαγιονείς ύφαλοι που προστατεύονται από την οδηγία για τα habitat και υπάρχουν και άλλα είδη ε, χελώνες λοιπά οι οποίες καλύπτονται από αυτή την οδηγία για την προστασία. Επίσης έχουμε και για τα κοιτόδη, έχουμε 35% της παρουσίας του, των κοιτοδών. Ε, εδώ έχουμε ας πούμε το ρινοδέλφινο, που και αυτό προστατεύεται από την οδηγία για το Habitat. Έχουμε επίσης ε, και άλλες άλλα είδη φάλαινος όπως η ριχοφάλαινα, φυστηρίδε κτλ. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό η μελέτη περιοδικών επιπτώσεων της τρεψολ ε, να πούμε ότι έχει πολλά σημεία που είναι αφανή, ε, ασαφή, χωρίς διαφάνεια και χρησιμοποίησαν για την μελέτη περιοδικών επιπτώσεων πολύ παλιά φιλολογία και δεν λάβα υπόψη τους νέα ε, σημεία από την επιστημονική φιλολογία που μιλούν για κίνδυνο για τα κοιτόδη ακριβώς στις περιοχές όπου προβλέπονται να γίνουν οι εξορίξεις. Είχαμε παρόμοια παραδείγματα στον κόλπο του Μεξικού όπου οι παλμοί, οι σεισμικοί παλμοί έβλαψαν ε, τις φυσιτηρίδες και αυτό αφορά ακριβώς την φύση των ε, κυμάτων του ήχου. Άλλο ένα σημαντικό στοιχείο είναι η χημική τοξικότητα από την λάσπη δριάτρησης. Λέει η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ότι έχουν γίνει μελέτες 500 μέτρα γύρω από τα σημεία εξόριξης, ενώ η επιστημονική φιλολογία λέει ότι αυτές οι περιοχές πρέπει να είναι μεταξύ 5 και 90 χιλιόμετρων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό επειδή αυτά, αυτές οι λάσπες ακριβώς ε, διάτρησης έχουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις στην σπονδυλωτή πανίδα και αφορά βεβαίω όλου του υδρογονάθρακε που προβλέπεται να εξορεχθούν. Το τρίτο μεγάλο λάθο ήταν η υποτίμηση των κινδύνων ή των ενδεχόμενων κινδύνων αυτέ τι δράσει στο Deepwater Horizon, το οποίο ήταν μια πλατφόρμα εξόρυξη, η οποία βρισκόταν σε παρόμοια βάθη με αυτό το σχέδιο της Repsol. Είχαμε ε, πλούμιο από υδρογονάθρακες και ε, είχαμε ότι για τα Κανάρια έχουμε μαροδέλφινα, ριχοφάλαινες και που ζουν στα Κανάρια συνέχεια όλο το χρόνο. Επίσης, λέει το Υπουργείο Βιομηχανίας της Ισπανίας ότι η μελέτη, η μελέτη περιβαλλοντικών επιδόσεων της Ρεψόλ είχε υποτιμήσει το ενδεχόμενο ε, πετρελοκυλίδα σε αυτές τις περιοχές. Βλέπετε εδώ λοιπόν στους ε, χάρτες ε, της Ρεψόλ ότι εδώ σε περίπτωση που υπάρχει πετρολοκυλίδα, υπάρχει διαρροή, θα καλύψει ένα πολύ μεγάλο τμήμα του Του αρχιπελάγους. Έχουμε θαλάσσια πανίδα, δελφίνια που ζουν σε αυτές τις περιοχές εδώ και πολλά χρόνια. Είδαμε μετά τον κόλπο του Μεξικού και την πετρολοκυλίδα εκεί ότι η υγεία τους ε, δέχτηκε σοβαρό πλήγμα. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. <clears throat> κοιτάξτε, δεν έχουμε πολύ χρόνο, γι' αυτό πρέπει να δώσω το λόγο αμέσως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ντάνιες Φερνάντες Γκόμες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να πω ότι εδώ εκπροσωπώ τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Γι' αυτό λοιπόν εγώ θα περιοριστώ στην παρέμβασή μου στις ε, μελέτες που η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος έχει κάνει σε σχέση με την ε, ε, μη σωστή εφαρμογή του περιβαλλοντικού δικαίου της Ένωσης. Θα ήθελα να δώσω το λόγο αμέσως στον κύριο Λίκμεν, τον συνάδελφό μου, ε, από την Γενική Διεύθυνση Ενέργειας ε, έτσι ώστε να δώσει τα ε, συμπεράσματα τα οποία απορρέουν από την μελέτη του θέματος. και σε προηγούμενες περιπτώσεις ενημερώσαμε την Επιτροπή Αναφορών ότι έχοντας ε, λάβει ε, τα διάφορα παράπονα πούμε των ε, αναφερομένων προσπαθήσαμε να διευκρινίσουμε εάν εφαρμόζεται σωστά το κοινοτικό δίκαιο όσον αφορά το περιβάλλον από πλευράς των Ισπανικών αρχών. Πληροφορήσαμε επίσης την Επιτροπή Αναφορών ότι ε, όταν θα είχαμε τις πληροφορίες από τις Ισπανικές Αρχές θα αναλύαμε τις πληροφορίες αυτές. Ε, έχοντας πράξει με τον τρόπο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ε, κατέληξε στο ότι δεν μπορεί να προσδιορίσει παραβίαση του κοινοτικού ε, δικαίου. Αυτή τη στιγμή δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η διαδικασία περιβαλλοντικού αντικτύπου και επίσης δεν έχει δοθεί ακόμα οποιαδήποτε άδεια. Εν τω μεταξύ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε πρόσβαση ε, σε ε, ε, πληροφορίες όσον αφορά τις, την ανάλυση αντικτύπου και όσον αφορά την αδειοδότηση ε, η οποία όμως δεν τροποποιεί τις, ε, τα αρχικά συμπεράσματα της Κομισιόν. Επίσης θα θέλαμε να σας πούμε ότι εντωμεταξύ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει ε, πολλές προσφυγές οι οποίες προκαλούν μια σειρά ερωτημάτων μεταξύ των οποίων και αυτά τα οποία παρουσίασαν οι αναφέροντες εδώ ε, όλα τα ερωτήματα των, τα, οποία έχουν φτάσει στην Κομισιόν αναλύονται. Δεν, έχουν, δεν έχει ακόμα όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκληρώσει την ανάλυση. Όταν θα έχει ολοκληρώσει την ανάλυση των παραπώνων ε, αυτών το, και των ετοιμάτων αυτών, ε, τότε θα δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενώπιον της Επιτροπής Αναφορών τα συμπεράσματά της. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λίγμαν από το τμήμα της ενέργειας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εκπροσωπώ τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας και βεβαίως είχαμε πολλές αναφορές και διαμαρτυρίες για παραβιάσεις της οδηγίας του 1994 που αφορά τις άδειες για την εκμετάλλευση, την εξόρυξη, την έρευνα καταρχήν, την εκμετάλλευση και την εξόρυξη υδρογων ανθράκων. Οι άδειες αυτές πρέπει να δίδονται με μια δίκαιη διαδικασία χωρίς διακρίσεις και βεβαίως ε, όλοι πρέπει να έχουν ίση πρόσβαση σε αυτές τις άδειες εκμετάλλευσης με βάση αντικειμενικά κριτήρια. Ελέγξαμε λοιπόν τις προσφυγές που έφτασαν μέχρι την δική μας ε, Γενική Διεύθυνση από κοινού με τις ε, Ισπανικές αρχές. Τουλάχιστον πρέπει να σας πω ότι αυτές τις οποίες εμείς ελέγξαμε δεν ε, διαπιστώσαμε καμία παραβίαση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Αυτό μπορώ να σας πω εγώ, τουλάχιστον από τη δική μας πλευρά, αυτό έχουμε διαπιστώσει. Okay, now... Εντάξει. Μπορούμε λοιπόν να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Ο κύριος Λόπες Αγκιάρα. Πρώτη ευχαριστώ. Είμαι εδώ εκπροσωπώντας τους σοσιαλιστές, την ομάδα τους και για να εκφράσω την υποστήριξή μας στην αναφορά που ακούσαμε τώρα ζωντανά. Υποδεχόμαστε λοιπόν εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών μη κυβερνικών οργανώσεων και πολιτών που ενδιαφέρονται για κάποιο ζήτημα το οποίο αφορά τις αρμοδιότητες της Ένωσης. Το κάναμε στις 21 του Γενάρη και πάλι οι σοσιαλιστές υποστηρίξαμε τους αναφερόμενους που προέρχονται από μη κυβερνικέ οργανώσεις, από οργανώσεις πολιτών, από περιβαλλοντικές οργανώσεις που βρισκόνταν σε μια μόνιμη κινητοποίηση υπέρ μιας θαλάσσιας ζώνης που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη και έτσι έχει ανακηρυχθεί από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό για να προσπιστεί επίση και το κοινωτικό δίκαιο. Όχι μόνο δηλαδή οι οδηγίες οι οποίες ακριβώς ρυθμίζουν την εξόριξη δρομοναθράκων αλλά και την οδηγία που αφορά τα άπειτα τους βιοτόπους του 92 που αναφέρθηκε εδώ. γιατί αυτή η πτυχή ακριβώς της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας θίγεται εδώ. Σχετικά δηλαδή με την προστασία πανίδας μιας ιδιαίτερης περιοχής που χαρακτηρίζεται από την μεγάλη παρουσία κοιτοδών σε μεγάλη συγκέντρωση παγκοσμία. 35% λοιπόν, όπως ακούσαμε από διάφορα κοιτοειδή βρίσκονται εδώ σε αυτή την περιοχή. Από τα 84 που ήδη και το εδώ που έχουν καταγραφεί παγκοσμίω, πολλά από αυτά βρίσκονται εδώ. Και αναφέρεται εξάλλου και στην ε, επιστημονική έκθεση που αναφέρθηκε και που έχουν προβάλλει και ακαδημαϊκές και επιστημονικές οργανώσεις που ασχολούνται με την προστασία των κοιτοειδών και των σπονδυλωτών στην περιοχή αυτή η οποία, τα οποία επιστημονικά στοιχεία αναφέρουν ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος από τις σεισμικές δραστηριότητες που αφορούν τις εξορίξεις. Η υποτίμηση του βαθμού τοξικότητας της λάσπης διάτρησης και το ενδεχόμενο πετρελαιοκελίδας γιατί όλοι θυμόμαστε τα πολύ σοβαρά ατυχήματα του κόλπου του Μεξικού, το Deepwater Horizon το 2010, που πέρασαν στην παγκόσμια ιστορία καταστροφών λόγω έλλειψης σωστού ελέγχου και των καταστρεπτικών επιπτώσεων που έχουν αυτές οι διαρροές όχι μόνο στο περιβάλλον αλλά και στην υγεία των ανθρώπων σε μόνιμη βάση. Εδώ λοιπόν ακούστηκαν στοιχεία σε σχέση με την ασυμβατότητα μεταξύ αυτών που πρόσφατα ήταν Υπουργοί Γεωργίας και Περιβάλλοντος της Ισπανίας για την ε, άμεση συμμετοχή τους σε εταιρείε πετρελαίου και μεταφοράς πετρελαίου. Να πω κάτι σημαντικό και το εξετάσαμε κατά τη διάρκεια της ακρόασης του υποψηφίου επιτρόπου. Οι εκθέσεις που προέρχονται από την, από κυβέρνηση της Ισπανίας, οι εκθέσεις αυτές υπόκεινται στις επιχειρηματικές στρατηγικές της, της Γιατί άλλαξαν τη διαμόρφωση του κοινοτικού, του ενωσιακού συμφέροντος και της πρόσπισης τους και έγιναν αλλαγές σοβαρές στις αδειοδοτήσεις το 2012 και άλλαξαν, άλλαξαν ακριβώς την περίμετρο προστασίας που απορρέει από το κοινοτικό ε, δίκαιο και αφορά συγκεκριμένα είδη. Υπόκεινται λοιπόν υπόκεινται τα στοιχεία που αφορούν την περίμετρο προστασίας στις επιθυμίες της Δεψόρ και όχι στις επιταγές της προσταγές προστασίας της κοινοτικής νομοθεσίας. Ξέρουμε λοιπόν και ακούσαμε τις επιπτώσεις σε αυτά τα είδη, τα θαλάσσια, από το, από το ενδεχόμενο εξορίξεων. Και ακούσαμε επίσης ότι μειώθηκε η περίμετρος οποία, την οποία συμβουλεύουν να εφαρμόζεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και έγινε σύμφωνη με τις επιθυμίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και της Ρεψόλ. Εδώ λοιπόν κυριαρχείται το δημόσιο συμφέρον από το ιδιωτικό, από την επιχείρηση αυτή τη Ρεψόλ. Υπήρχαν λοιπόν διαδηλώσει και κινητοποίηση των πολιτών των Καναριών νησιών και των τοπικών αρχών και τη τοπική κυβέρνηση. Είναι λοιπόν σημαντικό το Κοινοβούλιο να κάνει εδώ δουλειά σημαντική στην Επιτροπή Αναφορών, να κρατήσει ανοιχτή την αναφορά και να ζητήσει οι αναφερόμενοι να γίνουν δεκτοί με τα απαραίτητα συμπληρωματικά επιστημονικά στοιχεία από την Κομισιόν και την ε, Υπηρεσία για τα Περιβαλλοντικά Ζητήματα. Εμείς λοιπόν οι σοσιαλιστέ είμαστε υπέρ του να παραμείνει αυτή η αναφορά. Λοιπόν, ήσασταν πρόεδρος της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, δικό μου προέδρο. Ήθελα να σα διακόψω, αλλά δεν τόλμησα. Λοιπόν, με μεγάλη χαρά δίνω τον λόγο στην κυρία Λίπα, ε, Ριβάσο, αλλά μην μιλήσετε τόσο πολύ κι εσείς. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να μιλήσω λιγότερο. Να σας πω ότι το ίδιο πρόβλημα είχαμε και στην Μεσόγειο δίπλα στα νησιά Πορκρόλ και Πορκρό. Το λέω απλώς για να δώσω λίγη ελπίδα στα νησιά σας. Αν κινητοποιηθούν όλοι, μπορεί η κυβέρνηση να μην δώσει άδεια. Εμείς αυτό το πετύχαμε. Όταν είδα αυτό το θέμα, και εδώ αναφέρομαι στην Επιτροπή, κάνω έκκληση προς την Επιτροπή, η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, δεν, ε, πρέπει να, δεν, δεν μπορώ να σας πω ότι με εντυπωσιάσατε, γιατί πραγματικά δεν υπορασπίζεστε τα συμφέροντα που πρέπει. Μιλάτε για τον περιορισμό περιμέτρου, δεν στηρίζετε τις οδηγίες για τα πτηνά, για τα οικοσυστήματα. Λέτε ότι ουσιαστικά δεν πρόκειται για αυτό το θέμα. Το θέμα μας είναι οι υδρογονάνθρακες. Αλλά έχω την εντύπωση ότι η γενική σας διεύθυνση καταρχήν θα πρέπει όταν έγινε η μελέτη Ρεψόλ που από ό,τι βλέπουμε έγινε σε χρόνο ρεκόρ 40 ημέρες να υπάρξει μια πολύ πιο αποτελεσματική μελέτη που να λάβει υπόψη της το σύνολο των πτυχών του προβλήματος. Αν δεν το ζητείτε εσείς, ποιος θα το κάνει. Έχουμε τον κύριο Κανιέτε, ο οποίος θα γίνει επίτροπος αρμόδιος για θέματα ενέργειας και κλίματος, ο οποίος ήταν υπουργός περιβάλλοντος ο οποίος συμμετείχε σε αυτήν τη διαδικασία διοδότησης. Ήταν συνένοχος. Γιατί υπάρχει θέμα σύγκρουσης συμφερόντων, ήταν ε, μέτοχος ε, σε αυτήν την πετρελαϊκή. Τι να σας πω, αυτός είχε πει να αυξηθεί η περίμετρος. Τουλάχιστον να ξέρουμε πόσες ε, έρευνες και εξορίξεις θα γίνουν. Οι Ευρωπαίοι πολίτες, το είδατε από τις εκλογές, περιμένουν να προστατευθούν από την Ευρώπη. Και όχι μόνο στις Κανάριες νήσους και στην Πολωνία, παντού ισχύει αυτό. Αν δεν είμαστε απαιτητικοί όσον αφορά την πρόσβαση της πληροφορίας στην προστασία του περιβάλλοντος, τι κάνουμε. Αν υπάρξει κοιλίδα παραδείγματο χάρη αύριο. Τι μπορούμε να κάνουμε, τίποτα. Και ξέρετε πολύ καλά όσον αφορά τη σύμβαση στην ότι αυτό δεν πλήττει μόνο την Ισπανία αλλά και όλες τις ακτές, τις γαλλικές και άλλες, ανάλογα με το πόσο μεγάλη θα είναι η κοιλίδα. Άρα το θέμα είναι ευρωπαϊκό, δεν είναι εθνικό. Ζητώ λοιπόν η Επιτροπή να ζητήσει μια εναλλακτική μελέτη πιο σημαντική η οποία να λάβει υπόψη της όλα αυτά τα στοιχεία που σήμερα λείπουν από την πρώτη μελέτη της ε, Ρεψόλ και βεβαίως να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχει ευρωπαϊκή διάσταση και ότι εδώ πρέπει να αναφερθούμε σε περισσότερες οδηγίες αν δεν κάνετε τίποτα, βλέπετε ότι οι διεθνείς όμιλοι, οι οποίοι θέλουν να απεικοδομήσουν την Ευρώπη, θα οδηγήσουν τους Ευρωπαίους πολίτες στο να είναι ακόμα πιο δύσπιστοι προς την Ευρώπη. Βλέπετε επίσης ότι και το 2015 θα δοθούν νέες άδειες, συνεχίζουμε δηλαδή να ψάχνουμε για υδρογονάδρακες, να γίνονται εκμεταλλεύσεις, να γίνονται εξορίξεις, ενώ εμείς δίνουμε έμφαση και θέλουμε να στοχεύσουμε περισσότερο τις εναλλακτικέ πηγές ενέργειας. Πρόεδρος, έχω τέσσερις ομιλητές στον κατάλογο. Ήδη θα έπρεπε να είχαμε τελειώσει. Η κυρία Βαλίνα, ο Σεμπάγιος, Σεμπάστα και Μάρτα. Ευχαριστώ πολύ πολλά υπόθηκαν, γι' αυτό θα προσπαθήσω να μην με ακρηγορήσω, γιατί νομίζω ότι ε, όλα τα είπαμε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω και τους αναφέροντες ε, και όλα τα κινήματα τα οποία έχουν ξεκινήσει από τα Κανάρια νησιά, γιατί υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση για το πρόβλημα, για το πρόγραμμα αυτό ε, και για, τα, για τους αντικτύπους. Τα πράγματα δεν είναι απλά. Πρέπει οπωσδήποτε να μελετήσουμε αναλύσουμε σε βάθος εάν και κατά πόσον και σε ποιο βαθμό μάλλον έχουν παραβιαστεί κάποιες οδηγίες. Δεν αρκεί να δούμε κάποια ε, γενικά στοιχεία. Θα πρέπει να δούμε και το σορευτικό αποτέλεσμα που θα έχουν αυτές οι εξορίξεις. Αυτή τη στιγμή ε, δεν, ε, δεν εφαρμόζεται και η οδηγία για την πρόσβαση του κοινού στην πληροφόρηση. Δεν λαμβάνονται υπόψη τα προβλήματα λόγω των σεισμικών δονήσεων που θα προκληθούν ε, δεν λαμβάνεται υπόψη το ενδεχόμενο να παραμείνουν 300.000 άνθρωποι οι κάτοικοι του Λανθαρότε χωρίς πόσιμο νερό. Επίσης ε, δεν γίνεται λόγος για την παραβίαση της οδηγίας του 2004 ε, και όσον αφορά το σεβασμό των χρονικών περιθωρίων επίσης δεν έχουν ληφθεί υπόψη και επίσης θα πρέπει να δούμε εάν και κατά πόσον ένας υπουργός ο οποίος έχει συμφέροντα σε πετρελαϊκή ευρωπαϊκές εταιρείες είναι αυτός ο οποίος έδωσε το πράσινο φως για αυτό το πρόγραμμα εδώ. Υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Ε, θα πρέπει να ε, ε, τα δούμε όλα αυτά και επίσης θα πρέπει να τοποθετηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μονάχα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όχι μονάχα στα, στα επιστημονικά στοιχεία τα οποία έχει δώσει η Ισπανική κυβέρνηση αλλά και αυτά που έχουν δώσει έγκριτες επιστημονικές οργανώσεις. Ευχαριστώ πολύ. Το Πρόεδρε. Θα μιλήσω ισπανικά εδώ. Δεν διάβασα την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Διάβασα όμως πολλές μελέτες αντίστοιχες στα Κανάρια τα τελευταία χρόνια, γιατί εκεί δούλευα. Και από ό,τι βλέπω, υπάρχουν πολλές ελλείψεις, πολλά κενά, όπως και σε αυτήν την περίπτωση. Κάτι το οποίο βλέπουμε ξεκάθαρα παρόλο που διάβασα μόνο την περίληψη είναι ότι υπάρχει ένα κενό μεταξύ B και δήλωσης B. Και αυτό είναι κάτι το οποίο η Κομισιόν θα πρέπει να λάβει υπόψη της και να εξετάσει. Πρέπει να υπάρχει ένα πρωτόκολλο το οποίο συνοδεύει τις B και λέει ότι η ζώνη αποκλεισμού θα πρέπει να καθορίζεται από ειδικού, από εμπειρογνώμες. Αυτό όμως στην πράξη δεν ισχύει. Και αυτό είναι ένα από τα προβλήματα. Δεν έχουμε μόνο να κάνουμε μόνο με την ΠΕ, η οποία αμφισβητείται, η οποία δεν έχει γίνει από επιστήμονες, αλλά από αυτούς που θα κάνουν το έργο, τους εργολάβους. Και κάτι άλλο. Στα Κανάρια υπόθηκε ότι υπάρχει μεγάλη αντίδραση για το σχέδιο αυτό, όπως και για άλλα τεράστια σχέδια και προγράμματα που προγραμματίζονται για τα νησιά. Ο κόσμος βγαίνει στους δρόμους. Οπότε δεν αρκεί μόνο να το κάνει η κυβέρνηση αυτό. Η απόφαση πρόκειται από την κυβέρνηση της Ισπανίας. Συμφωνώ με αυτούς που είπαν εδώ ότι υπάρχει εδώ σύγκρουση συμφερόντα, αντικρώμενα συμφέροντα. Αυτό δεν κρύβεται και πριν λίγα χρόνια συζητούσαμε τον πρόεδρο του τοπικού κοινοβουλίου και μου ζήτησε βοήθεια στη, από μένα, βοήθεια από και από την κυρία Σέρλινγκ, ε, προηγούμενη ευρωβουλευτή στην οποία εργαζόμουν, ώστε να θέσουμε τέλος σε αυτά τα σχέδια εξόριξης. Δεν έχουμε να κάνουμε μόνο αυτό το σχέδιο, αλλά και άλλα σχέδια που αφορούν ε, τις ακτές των Καναρίων νησιών. Και τα Κανάρια ζουν ακριβώς από τον τουρισμό πολλοί Σουηδοί μεταξύ αυτών. Αν λοιπόν υλοποιηθούν αυτά τα σχέδια, τι θα γίνει με την οικονομία των Καναρίων και με την κοινωνία. Αυτό δεν αναφέρεται. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπε ο κ. Σαγγελάρ, ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε την αναφορά αυτή και να την αφήσουμε ανοιχτή. Είναι σημαντικό λοιπόν η Κομισιόν να εξετάσει τα επιστημονικά στοιχεία που θα προέρχονται από τους επιστήμονες που θα λάβουμε προσεχώς και κάτι άλλο που πιστεύω ότι είναι επίσης σημαντικό η Κομισιόν να μην πάει μόνο στη Μαδρίτη να ρωτήσει και να ζητήσει στοιχεία για αυτή την υπόθεση αλλά να πάει και αλλού να πάει ας πούμε στα Κανάρια και να μιλήσει με τον κόσμο οι οποίοι ξέρουν τι, τι συμβαίνει στις ακτές τους και όχι το Υπουργείο στη Μαδρίτη. Εγώ λοιπόν συμφωνώ απόλυτα με τις αμφορές αυτές, τις στηρίζω και θα ήθελα να ρωτήσω επί τη ευκαιρία και την Κομισιόν να μου πει αν έχει πάει στα Κανάρια με τον κόσμο ή αν έχει πάει μόνο στην Μαδρίτη. Αν έχει πάει μόνο στη Μαδρίτη, το να πάει και στα Κανάρια μιλήσει με τον κόσμο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας πω δεν πρόκειται για ένα θέμα που αφορά την Ισπανία ή τις Κανάρες νήσους. Πρόκειται για μια αναφορά που λαμβάνει υπόψη της την απόφαση της ε, Ισπανικής κυβέρνησης και είναι μια αντιευρωπαϊκή απόφαση κατά της περιβαλλοντολογικής νομοθεσίας που είναι η καλύτερη στον κόσμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, είναι κατά της ευρωπαϊκής πολιτικής σε θέματα ενέργειας που είναι υπέρ του καθαρού βιώσιμου μοντέλου ενέργειας. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι ο κύριος Κανιέτε, πρώην υπουργό Περιβάλλοντος, ήταν μέτοχος πετρελαϊκής ε, εταιρεία συγκεκριμένη αυτής που εμπλέκεται σε αυτή την υπόθεση. Είναι λοιπόν κάτι που δεν μπορούμε να το αφήσουμε χωρίς να διαμαρτυρηθούμε, γιατί εδώ βλέπουμε ότι και σε άλλα μέρη μπορεί να γίνει το ίδιο όσον αφορά τις άδειε στην Ισλανδία και αλλού στην Μεσόγειο. Αναρωτιέμαι λοιπόν και αναρωτιέμαι εδώ μπροστά σας στην Επιτροπή αν η Ευρώπη μπορεί να αφήνει τέτοιες αποφάσεις χωρίς να αντιδρά που παραβιάζουν τις περιβαλλοντικές μας αξίες. Είναι καθήκον μας να αντιδράσουμε και θεωρώ ότι οι πολίτες των νησιών, των Κανάριων νησιών, έχουν πάρει μια πολύ συγκεκριμένη θέση κατά αυτής της στάσης. Η Ευρώπη πρέπει να τους ακούσει, διότι οι άνθρωποι αυτοί αυτή τη στιγμή έχουν ξεκινήσει έναν αγώνα στο όνομα όλων μας. Και πολύ φοβάμαι ότι στο μέλλον θα υπάρχουν πολλά παρόμοια παράνομα σχέδια σε όλη την Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Ο τελευταίος ομιλητής είναι ο κύριος Μάτρεφ. Εγώ δεν είμαι πρόεδρος της ΛΥΜΠΕ, είμαι της Επιτροπής Αλίας, γι' αυτό μην μου βαρέσετε το σφυράκι αμέσω. Λοιπόν, για μία ακόμα φορά, όπως ε, ακούσαμε αυτό το πρόβλημα, δεν είναι η πρώτη φορά και πάντα ακούμε την ίδια απάντηση. Ε, εν περιπτώσει, θα ήθελα να θυμίσω ε, τι πρέπει να κάνει η Επιτροπή Αναφορών. Αυτό που πρέπει να κάνει είναι να ε, προωθήσει κάποιες αναφορέ. Ε, για τις ε, οποίες είναι σαφές ότι κάποιες αδειοδοτήσεις για εξόριξη υδρογονανθράκων παραβιάζουν συγκεκριμένες, ε, ε, συγκεκριμένες ενωσιακές ε, ρυθμίσεις ή νομοθεσίες. Εμείς δεν είμαστε εδώ για να δούμε και να συζητήσουμε για το εάν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων ή ακόμα λιγότερο βέβαια δεν είμαστε εδώ για να κατηγορήσουμε κάποιους. Υπάρχουν τα δικαστήρια για αυτές τις δουλειές. πρέπει να δούμε εάν αυτές οι αναφορές έχουν έννοια, έχουν περιεχόμενο και αναφέρονται σε κάποια παραβίαση κοινοτικού δικαίου. θα αναφερθώ θα αναφερθώ στο εξή. Στις 27 Νοεμβρίου του 2012, στις 19 Δοδεκάτου του 2013, ο επίτροπο Ποτόνικ ε, το 2014 έδωσε απάντηση σε μία ερώτηση βουλευτή ε, και είπε ότι η παραβίαση της, ε, της περιβαλλοντικής δικαιοσύνης, της νομοθεσίας δεν έχει υπάρξει. Επίσης, στι 29 Σεπτεμβρίου, πριν από μερικέ μέρες, το 2014, Επίσης είχαμε μία απάντηση. Αυτοί έχουν αποδομήσει όλα τα επιχειρήματα τα οποία αναφέρονται σε τούτες εδώ τις ε, ε, αναφορές. Δεν υπάρχει προδήλωση οποιαδήποτε παραβίαση από πλευράς της Ισπανικής κυβερνήσης. Ε, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω των δύο γενικών της διευθύνσεων το ίδιο έχει αναφέρει. Απ' την άλλη πλευρά το Ανώτατο Δικαστήριο με τελευταία απόφαση της 12ης Ιουνίου του 2014 έχει αποδομήσει ε, σημείο προς σημείο όλες τις διεκδικήσεις. Δεν μπορούμε να, ε, να δούμε εδώ τίποτα καινούριο. Δεν υπάρχει τίποτα νέο, καμία, κανένα καινούριο στοιχείο. Έχει γίνει ε, μια θεσμική ε, ε, και μια κοινωνική ανακοίνηση, ναι, είναι γεγονός. Υπάρχουν στοιχεία, υπάρχουν αποφάσεις οι οποίες κάνουν περισσότερο θόρυβο, προκαλούν περισσότερο θόρυβο, άλλες λιγότερο. Αυτό είναι αλήθεια. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχει η κυβέρνηση των Καναρίων που αποτελείται από τους σοσιαλιστές και από τους εθνικιστές των Καναρίων νήσων. Αυτή είναι κατά των εξορίξεων. και ε, ε, αναφέρουν ότι και έλεγε ο Γενικός Γραμματέας του Σοσιαλιστικού Κόμματος, ο οποίος είναι τώρα αντιπρόεδρος στην κυβέρνηση των Καναρίων, έλεγε πριν από λίγο καιρό, ε, εάν γίνουν αυτές οι εξορίξεις τότε θα υποστεί πλήγμα και ο τουρισμός και το περιβάλλον. Ε, και ότι εάν ε, υπάρχει όμως και η αντίθετη άποψη, την οποία έχουν εκφράσει επίσης έγκριτοι ομιλητές, οι οποίοι λένε ότι μόνο πλεονεκτήματα μπορούν να υπάρξουν σε περιπτώσεις ε, ε, εξορίξεων πετρελαϊκών στα Κανάρια ε, και αυτό το έχει πει ο ε, παλαιός ηγέτης των σοσιαλιστών στα Κανάρια που είναι τώρα στην κυβέρνηση των Καναρίων ε, νήσων. Ε, επίσης και ο τέος πρόεδρος των Καναρίων έλεγε παλιότερα δεν υπάρχει καμία δυνατότητα σε καμία χώρα του, του, κόσμου εάν υπάρχουν πιθανότητες εξέβρεσης πετρελαίου να μην προχωρήσει σε εξόριξη. Λοιπόν, πότε λένε έχουν δίκιο όταν λένε το ένα ή όταν λένε το άλλο. Πότε λένε αλήθεια, πότε λένε ψέματα οι ίδιοι άνθρωποι που εκπροσωπούν τους ίδιους φορείς. Επίσης αυτό που είναι σαφές είναι ότι ε, αυτές ε, οι αναφορές ε, περιλαμβάνουν στοιχεία τα οποία δεν είναι σωστά ή είναι ασαφή. Αναφέρεται στην, στην απόσταση που θα έχουν αυτές οι εξορίξεις από τις ακτές του Λανθαρότε ή από τις ε, ακτές ε, της Φουερτεβεντούρα Δεν έχουν δοθεί σωστά αυτά τα στοιχεία. Γίνεται λόγος επίσης για το βάθο των ε, υδάτων, ούτε τα στοιχεία αυτά όμως είναι σωστά. Εν πάση περιπτώσει εν κατακλείδη δεν υπάρχουν νέα στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται σε αυτές τις αναφορές. Επίσης ε, αναφέρονται και στοιχεία τα οποία δεν είναι ε, σωστά, ότι δεν υπήρξε δημόσια διαβούλευση, ότι δεν δόθηκε στη δημόσια διαβούλευση ο χρόνος που έπρεπε. Όχι, 45 μέρες πριν ξεκινήσει η δημόσια διαβούλευση είχε κοινοποιηθεί αυτή. Εν πάση περιπτώσει νομίζω άλλωστε ότι μερικοί δεν έχουν διαβάσει καλά τις μελέτες, γιατί η μελέτη που αναφέρουν ακριβώς λέει ε, ότι ότι ε, πέρα από την έγκριση των ε, προγραμμάτων ΛΙΚ ε, θεωρήθηκε ότι είχαν ολοκληρωθεί ήδη οι μελέτες περιβαλλοντικού αντικτύπου. Μα δεν είναι αυτό, δεν ισχύει όμως γιατί δεν είχαν εγκριθεί τα ΛΙΚ. Εν πάση περιπτώσει, σας λέω, δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να παραμείνουν ανοιχτές αυτές οι αναφορές, δεν έχουν τίποτα καινούριο. Επίσης, νομίζω, νομίζω ότι ε, σε αυτή την περίπτωση οι δηλώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι σαφέστατες. Οι αρμοδιότητες είναι σαφέστατες επίσης. Τα αιτήματα των αναφερομένων επίσης είναι σαφή. Οι απαντήσεις πρέπει να είναι εξίσου σαφές. Δεν νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να συνεχίσουμε να παίζουμε αυτό το κρυφτούλι ε, ε, για ένα θέμα το οποίο έχει ξεκαθαριστεί πλέον. Ε, εντάξει, μπορεί κάποιο να πει ότι είτε η Κομισιόν δεν είναι καλή, είτε ότι αυτά που λέει η Κομισιόν δεν είναι καλά γιατί δεν τις αρέσει. Απ' την άλλη πλευρά όταν ε, ε, τους δώσουν δίκιο θα πούνε «Α, τι εξαιρετική που είναι η τεχνική και οι, ε, οι μελέτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής». Νομίζω ότι εδώ έχουμε, πρέπει να σεβόμαστε την εργασία των ανθρώπων που αποτελούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, των εμπειρογνωμόνων που δουλεύουν για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. με σεβασμό βλέπουμε αυτά που έχουν ζητήσει οι αναφέροντες, αλλά δεν υπάρχει τίποτα καινούριο έτσι ώστε να συνεχίσουμε με, ανοιχτή την επιτρο... τις, ε, τις αναφορές αυτές. Νομίζω ότι τα υπόλοιπα ζητήματα θα πρέπει να λυθούν ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων, εάν και εφόσον προκύψουν τέτοια. Και εάν υπήρχε, εάν προέκυπτε κάποιο καινούριο στοιχείο, εάν αποκαλυφθεί κάτι νέο, τότε βεβαίω οποιαδήποτε στιγμή είμαστε στη διάθεση των αναφερομένων έτσι ώστε να υποβάλουν νέα αναφορά. Δεν είναι δυνατόν ε, ελήψη οποιοδήποτε αντικειμενικού λόγου να συνεχίσουμε να ασχολούμαστε με το ίδιο θέμα. ευχαριστώ πολύ. Πολλοί συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο. Δεν είναι δυνατόν να δώσουμε ε, το λόγο τώρα. 20 λεπτά έχουμε καθυστερήσει. Μαργκρίτα, ζητάς το λόγο. Λοιπόν, οι διερμηνείς έχουν δείξει πάρα πολύ μεγάλη ε, υπομονή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε όλοι πάρα πολύ κουρασμένοι και εμείς και εσείς. Βεβαίως καλό θα ήταν να ξαναδίναμε το λόγο στην Κομισιόν και στον ε, αναφέροντα, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Προτείνω λοιπόν το εξής. Η μόνη πρόταση ε, είναι η πρόταση του κυρίου Μάτο να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά όχι, όχι, δεν είπα αυτό. Εγώ είπα το αντίθετο. Εγώ είπα να κλείσει, να κλείσει η αναφορά και να ξανανοίξει εάν και εφόσον προκύψουν νέα στοιχεία. Yeah, exactly. I wanted to say exactly. Ακριβώς, ακριβώς το αντίθετο είπατε. Να κλείσουμε την αναφορά, αυτό προτείνατε. Όλοι οι άλλοι όμως είπαν να παραμείνει ανοιχτή. Άρα... Αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε σαν Επιτροπή Αναφορών είναι να στείλουμε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις νέες επιστημονικές μελέτες που διαθέτουμε και να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διευρύνουν τις έρευνές τους, τις μελέτες τους με αντικειμενικό τρόπο και να δουν αν υπάρχει κάτι καινούριο σε αυτά τα νέα στοιχεία και να υπάρξει και μια νέα αξιολόγηση που να βασίζεται στα νέα επιστημονικά στοιχεία. Νομίζω ότι η μεγάλη πλειοψηφία υποστηρίζει αυτήν την άποψη, περισσότεροι συνάδελφοι της Επιτροπής. Λοιπόν, ή κλείνουμε ή παραμένει ανοιχτή. Πρόεδρε, συμφωνώ με την πρότασή σας να λάβουμε δηλαδή όμως τις νέες ε, εκθέσεις τις επιστημονικές το ταχύτερο δυνατόν. Δεν έχω καμιά αντίρρηση να σταλούν στην Κομισιόν για να αξιολογηθούν. Ωραία. Τέλος της συνεδρίασης συμφωνούμε όλοι. Η επιστημονική αξιολόγηση, τα επιστημονικά δεδομένα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Σας ευχαριστώ πολύ.